Ehm, Καλημέρα αξιότιμοι συνάδελφοι. Σήμερα έχουμε πολύ φορτωμένη ημέρα. Τα πάνελ ε, βρίθουν εισηγητών. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, σας προτείνω να θετήσουμε την αδιάταξη διάταξη της σημερινής συνεδριάσεως όσα σε προτάφει. Και αν δεν έχετε αντιρρήσεις, σας προτείνω να εθετήσουμε και τα πρακτικά της συνεδριάσης 21ης Μαΐου που μας πέρασε όσα σας επροτάθη. Τέλος, να σας υπενθυμίσω, η συνεδρίαση των συντονιστών της ΚΡΙΜ θα γίνει και κλεισμένων των θυρών εδώ από τις 5 και 4 και μετά. Όπως σας έλεγα, αυτό το πρώτο τμήμα της συνάντησής μας, συνεδριά συνεδριάσεως μου, θα αφιερωθεί σε μια αξιολόγηση Τη εμβέλειας και τη συνέπεια του οργανωμένου εγκλήματος και των μαφιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πάνελ είναι πλούσιο από εισηγητές υψίστου επίπεδου που αντιπροσωπεύουν και εκπροσωπούν τις καλύτερες αρχές εθνικές και ευρωπαϊκές όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Σήμερα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις των επαϊόντων και Θεωρώ ότι είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό τη συνέχεια των εργασιών μου. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω ονόματι τη Επιτροπή, τον Δόκτωρα Κέστρερ, τον Γενικό Διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμηση τη Απάτη, Όλαφ. Πριν ακούσουμε τον κύριο Διευθυντή, σα προτείνω να διθώσουμε τη συζήτηση ε, όπω συνήθω δηλαδή, να δώσουμε το λόγο παρεθή στον Δόκτωρα Κέστρε για την παρουσίασή του. Ευθύ μετά, πρώτο γύρο ερωτήσεων θα ακολουθήσει για τους συντονιστές των ομάδων και μετά εκ νέου λόγο στον κύριο Διευθυντή και μετά αν έχουμε το χρόνο θα δώσουμε το λόγο στους άλλους ε, βουλευτές. Λοιπόν, ε, δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Διευθυντή. Καλημέρα, ευχαριστώ όλους σας. Θα κάνω σε μερικά λεπτά μια εισαγωγή και να δώσω κάποιες πληροφορίες και κάποιο μήνυμα αν θέλετε από την πλευρά μου να σας δώσω και μετά είμαι στη διάθεσή σας για μια συζήτηση που πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρουσα και για την υπηρεσία που εκπροσωπώ και τη θέση μου. Η Όλαφ λοιπόν, η υπηρεσία καταπολέμησης των απατών όπως γνωρίζετε είναι το, η μόνη υπηρεσία, η ερευνητική μόνη ερευνητική υπηρεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ε, άλλοι φορείς ευρωπαϊκοί στον τομέα της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης του εγκλήματος, αλλά καμία, κανένας από αυτούς τους φορείς δεν έχει εντολή ερευνητική εξυχνίασης. Αυτό μας επιτρέπει λοιπόν να επεξεργαστούμε κάτι που θα βασίζεται στη δική μας εμπειρία και θα ήθελα πρώτης και εντάχει να σας δώσω κάποια ιδέα σχετικά με αριθμητικά στοιχεία και να σας παραθέσω επίσης κάποιες προπτικές σχετικά με αυτά που κάνουμε. Εμείς λοιπόν αναλύσαμε όλες τις έρευνές μας που διενεργήθησαν την τελευταία διετία, τριετία, δύο χρόνια, ζητώ συγγνώμη, 2009-2010 για να είμαι ακριβής, είναι οι χρονιές όπου κάναμε στοχευμένη στατιστική ανάλυση για να δούμε πώς από αυτές τις υποθέσεις που ερευνήσαμε απατών ή αδικημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μπορούν με ασφάλεια να θεωρηθούν ότι έχουν διαπραχθεί από το οργανωμένο έγκλημα. Από 375 έρευνες που έκανε η υπηρεσία μας, και ολοκλήρωσε στη διετία που προανέφερα 35 υποθέσεις 10% πάνω κάτω των υποθέσεων σχετίζονται, σχετίζεται άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα. Η οικονομική συνέπεια τώρα των υποθέσεων αυτών. Από 375 έρευνες είδαμε ότι αφορούσαν 1 δις 700 εκατομμύρια ευρώ υποθέσεις. Το υπολόγισε αυτό η υπηρεσία μας. Αυτή είναι η ζημιά που ε, δημιουργήθηκε από τις απάτες και τη διαφθορά. Δηλαδή, από τις 275 αυτές υποθέσεις. Ποιος είναι ο αντίκτυπος, ο οικονομικός, αυτών των 35 ερευνών που σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα είναι 750 εκατομμύρια. Πάνω το 40% του γενικού, της γενικής οικονομικής ζημιάς δηλαδή. αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Η δική μας εμπειρία μας λέει κάτι. Μας αποδεικνύει κάτι που ίσως μπορούσαμε να το διστανθούμε, αλλά τώρα εδώ έχουμε τα στοιχεία. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι το 10% των ερευνών για το οργανωμένο έγκλημα, που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, αφορούσε υποθέσεις που ε, οι οικονομικέ συνέπειε αυτών των υποθέσεων είναι πάνω το 40% τη γενική οικονομική ζημία. Δηλαδή, τα αδικήματα που, τα εγκλήματα που ερευνήσαμε και σχετίζονται με το οργανωμένο έγκλημα ε, έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική συνέπεια κατά των συμφώνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να πούμε και με βάση την εμπειρία μας, την εμπειρία μας λέω, με τα εμπειρικά μας αυτά τα στοιχεία, ότι το οργανωμένο έγκλημα είναι το πιο επικίνδυνο, το πιο επιζήμιο οικονομικά όσον αφορά τα ευρωπαϊκά οικονομικά συμφέροντα. Τέσσερις φορές μεγαλύτερη ζημιά σε σύγκριση με τα άλλα είδη, είδη εγκληματικότητας. Όταν μιλάω για οργανωμένο έγκλημα, στην ανάλυση μας ήμασταν πολύ προσεκτικοί για να αποσταλήσαμε το οργανωμένο έγκλημα. Λάβαμε υπόψη τις έρευνες που έδιναν τη βεβαιότητα της εμπλοκής του οργανωμένου έγκληματος και βλέπουμε από την εμπειρία μας από αδικήματα και εγκλήματα που είχαν οικονομική, οικονομικό αντίκτυπο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπαμε λοιπόν και είδαμε ότι αυτά τα εγκλήματα και δραστηριότητε που εμπλέκεται το οργανωμένο έγκλημα πάνω απ' όλα είναι το λαθρεμπόριο το διεθνές, κυρίως λαθρεμπόριο σιγαρέτων. Εξαιρετικά επιζήμιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικός πόσο. Και το λαθρεμπόριο εν γέννη. Πέραν αυτού, βλέπουμε ότι ένα βασικό έγκλημα που είναι πολύ σημαντικό και συχνά συνοδεύει την εγκληματική δραστηριότητα. Το οργανωμένο είναι η διαφθορά, το φαινόμενο της διαφθοράς. Είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το οργανωμένο έγκλημα σε αυτού του είδους τα εγκλήματα. Και το λαθρεμπόριο. Και στο λαθρεμπόριο μάλλον. Λοιπόν, όσον αφορά αυτά τα στοιχεία, να προβάλλω και κάποιες σκέψεις και τι προοπτικές δημιουργούνται. Αυτά λοιπόν τα εγκλήματα εν γέννη που είναι επιζήμια για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πιο συγκεκριμένα τα δικήματα, τα εγκλήματα του οργανωμένου εγκλήματος, η πράξη του οργανωμένου εγκλήματος που λαμβάνουν χώρο εντός Ευρωπαϊκής Ενώσεως, σε επικρατείες, έχουν διεθνή υπερεθνική διάσταση, όλο αυξανόμενη. Όταν μιλάμε για αυτές τις πράξεις οργανωμένου εγκλήματος, αναφερόμαστε σε αυτέ που δημιουργούν ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα συμφέροντα τα οικονομικά και πολύ συχνά και όλο και περισσότερο αναφερόμαστε σε εγκλήματα που από τη φύση του έχουν υπερεθνική διάσταση. Εγώ κάθε φορά που έρχομαι στο Κοινοβούλιο σαν διευθυντή τη Όλαφ και βλέπω του δημοσιογράφου μετά με ρωτάνε ποια είναι η χώρα και χτε με ρωτούσαν δύο φορέ ποια είναι η χώρα μου λένε τη Ευρώπη που έχει περισσότερε απάτε. Και γιατί αυτή η χώρα και όχι άλλη. Και εγώ κάθε φορά του απαντάω ότι είναι δύσκολο να κάνεις εθνικές διαβαθμίσεις. Να κάνουμε, να κάνουμε πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, ένα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου στον φάτσα πάτες. Ο καθένας ε, κοιτάει τη χώρα του και τη γειτονική, λίγο πολύ. Η διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, επίσης, λόγω δραστηριοτήτων έχουν εδαφική μορφή και ρίζε και προέλευση, το ξέρουμε την Ιταλία, αλλά στις δραστηριότητε τους, που είναι επιζήμιες για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης, δεν γνωρίζουν όρια και σύνορα. Η διαφθορά μπορεί να λάβει χώρα σε, μια, σε ένα κράτος, αλλά χρειάζονται δύο πλευρές. Από τη μία πλευρά ο δημόσιο υπάλληλο που πληρώνεται και ίσω αυτό που πληρώνεται σε άλλη χώρα. Πληρώνονται τα χρήματα σε, άλλη, σε τρίτη χώρα στο διεθνές λαθρεμπόριο των τσιγάρων, παραδείγματο χάρη. Στατιστικά μα στοιχεία φαίνεται στο Βέλγιο ή στην Ιταλία. Διότι το πλοίο κατεσχέθη στην Ιταλία στο Βέλγιο, αλλά είναι ένα έγκλημα που έγινε, είναι Ιταλικό, είναι Βελγικό, είναι Γερμανικό, γιατί έφτασε το πλοίο στο Αμβούργο. Από ποια χώρα προέρχεται. Μιλάμε τώρα για οργανώσεις που μπορεί να έχουν συγκεκριμένη προέλευση και ρίζες, όμως δρούν εντό Ευρωπαϊκή Ενώσεω και στον κόσμο με έναν τρόπο που δεν συνδέεται με συγκεκριμένη χώρα. Οπότε, και αυτό είναι το μήνυμα τώρα, το ισχυρό μήνυμα που θέλω να σας δώσω. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που συχνά στρέφεται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενώσεω δεν μπορεί να λάβει χώρα μόνο σε εθνικό επίπεδο. Μόνο από, εθνικής, επιθυνικού επίπεδο αν γίνει ε, δημιουργείται ένας κίνδυνος αν γίνει αυτό. Να μην δούμε την εικόνα στο, τη γενικότερη. Να βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Και από πλευρά ερευνητική εθνική προσέγγιση δημιουργεί το κίνδυνο να μείνουν εκτός εστίασης ε, τα μεγαλύτερα κομμάτια του φαινόμενου. Μετά, στις έρευνες Οι εθνικές αποκλειστικά έρευνες και η χρήση διεθνών και ανάγκη χρήσης διεθνών επιχειρήσεων είναι ένα μειονέκτημα, είναι ένα όριο και δεν αρκεί για τη σωστή έρευνα. Ας πούμε το διεθνές ένταλμα των διεθνών έρευνων είναι ένα τα θετικά μέσα που ίσως είναι ανεπαρκή στα πλαίσια της ε, δικαστικής συνεργασίας. και είναι και ανεπαρκή και αργή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών και χρειάζονται εθνικές αρχές που ασχολούνται με εθνική μερική έρευνα, διαφορετική προσέγγιση, έρευνα του ίδιου ε, φαινομένου. Όποτε έχουμε ε, μια προσέγγιση καλλιδοσκοπίου και δύσκολο από αυτή την μερική οπτική γωνία, την τμηματική θεώρηση των πραγμάτων, να δημιουργηθεί μια σφαιρική προσέγγιση και αντιμετώπιση του κλιματικού φαινομένου. Τα μέσα λοιπόν που έχουμε είναι παραδοσιακά μέσα. Της δεκαετίας του, του, του, της εποχής του 1800, του 19ου αιώνα και είναι ανεπαρκή αυτά τα μέσα που ήταν των εθνικών κρατών να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο που είναι πολύ ευρύτερο και όσον αφορά την οικονομική του εμβέλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγα στην αρχή, διαθέτει ένα και μοναδικό ερευνητικό μέσο, ευρωπαϊκό και υπερεθνικό, την Όλαφ. Η Όλαφ όμως, να μην το ξεχνάμε, για να μην δημιουργούμε και αβάσιμες προσδοκίες, εξορισμού είναι ένα μέσο διοικητικής έρευνας. Δεν έχουμε εξουσίες δικαστικές, αρμοδιότητες. Και οι έρευνές μας μετά καταλήγουν στην εθνική δικαιοσύνη, στις εθνικές εισαγγελίες και πολλές υποθέσεις δεν ξέρουμε σε ποια ε, ε, εθνική υπηρεσία θα πρέπει να απευθυνθούμε όταν είναι υπερεθνικό το έγκλημα. Άρα χρειάζεται μετά να επαναληφθεί σε εθνικό επίπεδο η έρευνα στα πλαίσια εκείνης της δικαστικής τάξης της χώρας. Μεγάλο όφελος έχει όλα, γιατί επιτρέπει σφαιρική θεώρηση ευρωπαϊκή των πραγμάτων, ανακάλυψη, εξυχνίαση Ενό είδου, ενό τύπου ε, εγκλημάτων που σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να μην εντοπιστούν έχει αυτό το όφελος. Και μετά μπορεί να κινηθεί κανείς και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και εκτό Ευρώπη. Με πολύ μεγάλη ελευθερία. Διότι δεν δεσμευόμεθα, δεν ε, περιοριζόμαστε σε εθνική επικράτεια, αλλά μετά στι συνέπειε η έρευνά μα περιορίζεται στα αποτελέσματα, διότι θα πρέπει να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη την εθνική. Άρα ξαναρχίζει η όλη διαδικασία. Εγώ πιστεύω και κλείνω εδώ, εκφράζοντας ελπίδα, μήνυμα, πρόταση, πάρτε το όπως θέλετε, ότι αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι ερευνητική υπηρεσία ευρωπαϊκή, ε, βάση Όλαφ ε, και Eurojust, η οποία όμως να έχει την εξουσία στα πλαίσια των ερευνών τη να σκίσει άμεσα ποινική δίωξη, ποινική δράση κατά ε, ε, έναντι των εθνικών αρμοδίων δικαστικών οργάνων. Κάτι σαν την Όλαφ, αλλά που θα έχει το δικαίωμα παράλληλα να διενεργεί δικαστικές έρευνες, δικαστικού τύπου, και αυτή η υπηρεσία να έχει και τη δυνατότητα να ασκήσει ποινική δίωξη. Το Ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εισαγγελία που προβλέπεται από τη συνθήκη πιστεύω ότι είναι το πραγματικό εργαλείο που θα μας οδηγούσε σε ένα μεγάλο ποιοτικό άλμα και θα ήταν μεγάλη πρόοδος για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για αυτή την παρουσίασή σας, αλλά πάνω από όλα διότι εστιαστήκατε και επειδή υπογραμμίσατε κάποια βασικά σημεία των, ε, τα οποία θα συζητήσουμε εξάλλου. Θα δώσω το λόγο παρευθύς στους συντονιστές και εκείνους που αντικαθιστούν τους συντονιστές. Παρακαλώ να μιλήσετε μόνο ένα δίλεπτο για να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να μπορέσουν να μιλήσουν. Δίνω το λόγο στον κύριο Ντίας Δεμέιρα που αντικαθιστά τον κύριο Ματίου. Όχι λέει του ΕΛΚ. Όχι, δεν ζήτησα το λόγο κυρία Πρόεδρε. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τα όσα λέγει ο κύριος Κέσλερ, αλλά δεν ζήτησα το λόγο. Καλώς. Η κυρία Μπορσελίνο θέλει να μιλήσει. Και εγώ δεν ήθελα να μιλήσω τώρα, αλλά είναι σημαντικό το ότι ανοίγουμε με ένα όραμα σαφέστατο. Θα ήθελα να δοκιμάσω να συνοψίσω. Απλά. Ακούσαμε μια εξαντλητική αναφορά της Όλαφ, ο πλευράς του διευθυντού της. Ακούσαμε ποια είναι η οικονομική ζημιά που δημιουργεί η απάτη. Ζημιά για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρώπης οικονομική ζημία που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη διότι δεν είναι μόνο αυτό που αφαιρείται εντό εισαγωγικών από την νόμιμη οικονομία, από την υγιή οικονομία αλλά είναι και ένα πρόβλημα εικόνας. Πρόβλημα της μείωσης ας πούμε της εμπιστοσύνης. Από πλευράς εκείνων πλησιάζουν αυτού του είδους τις παραγωγές. Θα ήθελα να πω ότι τα συμπεράσματά σας κύριε Διευθύντα βλέπω ότι όλα Όλαφ όπως και τα άλλα ευρωπαϊκά μέσα είναι σαν έμβρια. Ε, εμπεριέχουν όλα τα αναγκαία και χρήσιμα στοιχεία για να μπορέσουν ε, να πετύχουν το στόχο τους αλλά σε κάποιο σημείο δεν μπορούν να ζήσουν με την ίδια, ζωή, την ίδια τους τη ζωή και να αναπτυχθούν διότι περιορίζονται και στριμώχνονται από τις διάφορες χώρες γενικά, με τις οποίες πρέπει να έρθουν σε επαφή όταν πρέπει να περάσουν τη δικαστική φάση. Σαν προληπτική φάση, διοικητική φάση, καλά πάντα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτό που χρειάζεται είναι μεγαλύτερο συντονισμός, συνεργασία, δυνατότητα ανταλλαγής, ανταλλαγών διότι το οργανωμένο έγκλημα έχει πολύ πιο προχωρημένα εργαλεία και πιο ελεύθερο είναι το οργανωμένο έγκλημα. Δεν χρειάζεται να συμμορφώνεται στις διάφορες νομοθεσίες των χωρών. Οπότε θα έλεγα ότι χρειάζεται να βάλουμε κάτω από μια κοινή αιγίδα, ίσως στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας, που να μην αφορά μόνο τη συνεργασία μεταξύ ξεχωριστών φορέων, αλλά να έχει κοινό φύλλο θα ήθελα να καταλάβω κατά πόσο αυτή είναι η σωστή ερμηνεία. Έχουμε ένα έμβριο που χρειάζεται να αναπτυχθεί για να γίνει κάτι ε, αυτόνομο και να μπορεί να αναπτυχθεί. Ευχαριστώ κυρία Μπορσελίνο. Ο κύριος Νιούτον Ντόν για την άλλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Διευθυντά, Ακρο ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Είναι σύντομος ο χρόνος, αλλά είμαι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να τα ξανασυζητήσουμε. Γνωρίζω ότι η Επιτροπή μας πρέπει να απευθύνει συστάσει για το πώς θα μπορούσε η Ένωση να βελτιωθεί. Εάν δεν μπούμε πάρα πολύ ξεκάθαρα τι θα πρέπει να κάνει η Ένωση, θα χάσουμε την ευκαιρία αυτή για 5-10 χρόνια υπενηχθήκατε ε, στην ομιλία σας και εγώ με μανία σημείωνα. Μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα χαρτί αργότερα, αν θέλετε και χωρίς το όνομά σας, γιατί ε, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι επικίνδυνο και επιλύει τη δουλειά σας. Αλλά τι χρειαζόμαστε στην Ευρώπη, ένα FBI, ποια είναι η δομή που θα πρέπει να έχουμε, εισαγγελέα θέλουμε, ε, το υπενηχθήκατε και αυτό. Μήπως χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά ποινικά δικαστήρια για να δικάζουμε αυτούς τους ανθρώπους, κυρώσεις τι κυρώσει φυλακέ. Υπάρχει ιεράρχηση των ε, πραγμάτων και θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια για τα δικά μας συμπεράσματα να μας πείτε τι κάνει η Ευρώπη και τι χρειάζεται η Ευρώπη σε ένα ιδανικό κόσμο για να πιέσουμε το χρόνο που θα κάνουμε την έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ. Και στάση για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, σας άκουσα, κύριε Κέσλερ ε, με μεγάλη προσοχή. Έχουμε ξανασυναντηθεί και στο παρελθόν. Ε, τονίζεται πάρα πολύ την εμπειρία που έχει ο Όλαφ στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο ε, σιγαρέτων. Και νομίζω ότι η Task Force λειτουργεί καλά γύρω από το λαθρεμπόριο καπνού και τσιγάρων. Θα μπορούσατε να, να μας πείτε ποια διδάγματα έχετε εξαγάγει από αυτή την εμπειρία σας. Πέρα από το γεγονός ότι καταπολεμάτε καλά και συντονίζετε καλά αυτή την προσπάθεια στο εσωτερικό της Όλαφ για το λαθρεμπόριο τσιγάρων, μπορείτε να βρείτε ποιες είναι οι ελλείψεις. Γιατί αυτό το είδος λαθρεμπορίου συνδέεται όλο και περισσότερο με άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Διαβάζω ότι υπάρχουν σπήρες που διακινούν ανθρώπους, όπλα, τσιγάρα και ξέρω τι άλλο. Ε, μπορείτε να μας δώσετε τη δική σας προσέγγιση ή μια εικόνα έτσι υποπτική. Για πόσα λεφτά μιλάμε στο λαθρεμπόριο των τσιγάρων, πόσα χρήματα χάνονται ε, από ε, το κρατικό κορβανά του κάθε κράτους μέλους, από τα έσοδα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τελική ανάλυση. Και σε ποια τάξη μεγέθους αυτό το είδος εγκληματικότητας ε, εκτιμάται από τις υπηρεσίες σας στην όλα αυτές τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ.

Αλλά ε, τι χρησιμοποιείται ως ορισμό ε, για να λέμε ποια είναι αυτά τα εγκλήματα και η απάτη. Μετά, ε, η απάτη σε ό,τι αφορά τα έσοδα της Ένωσης έχει αυξηθεί κατά την Όλαφ σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο έχει παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Τρίτον, όταν μιλούμε για λαθρεμπόριο και απάτη είναι πάρα πολύ θαλά τα νούμερα. Μας δώσετε κάποια στοιχεία, αλλά έχετε καθόλου εκτίμηση για το πόσο υψηλό είναι αυτό το ποσό που δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Και αυτό που προτείνεται με ΑΙ ως λύση είναι ενδεχομένω μια ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αλλά είναι αυτό μια δραστηριότητα εγκληματική μόνο στο εσωτερικό της Ένωσης. Ε, και στο εξωτερικό. Αναφερθήκατε σε 375 περιπτώσεις. Πόσες είναι στο εσωτερικό της Ένωσης και πόσες εκτός. Κύριε Διευθυντά, επίσης μας είπατε ότι υπάρχει θέμα δωροδοκίας, διαφθοράς. Αυτό πώς γίνεται. Ποιο στόχο έχουν να βγάλουν χρήματα για να μπορέσουν να δωροδοκίσουν κάποιους για να δούμε και πώς διακινείται αυτή η κατάσταση και πώς μπορεί να καταπολεμηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μιλώ εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Ε, λυπάμαι πάρα πολύ. Έχασα ε, την ε, ε, παρέμβασή σας τα περισσότερα, γιατί με καθυστέρησαν ε, πριν φτάσω εδώ. Μπορείτε να μας πείτε ιδιαίτερα κάτι για την παραχάραξη του ευρώ. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται Περικλής. Εργάζεται και ο κύριος Δεμέρα σε αυτή την κατεύθυνση και εγώ, ε, ακριβώς για την ε, καταπολέμηση και την πάταξη της παραχάραξης του ευρώ. Και θα ήθελα να μας πείτε τι φρονείτε σχετικά. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στον κύριο Κέσσα, τον κύριο Διευθυντή. Καλώς. Όπως σωστά υπόθηκε, ίσως χρειάζεται και μια δεύτερη συζήτηση, δεύτερος γύρος, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα, χρειάζεται μια ανάλυση εμβριθής. Με ρωτάτε τι χρειαζόμαστε. Αυτό ρωτήσατε και η κυρία Μπορσελίνο κατά κάποιο τρόπο ακολούθησε την ίδια προσέγγιση. Χρειαζόμαστε ένα θεσμό εργαλεία. Στην, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εργαλεία που να μπορούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση. Ε, πράγματα που μας λείπουν. Δεν έχουμε. Είναι πιο πολύ προχωρημένοι. Επιχειρηματικά. Είναι επαγγελματίε. Πιο προχωρημένοι αυτοί από μας πιο οργανωμένοι. Έχουμε εργαλεία που χρονολογούνται τουλάχιστον τον περασμένο αιώνα. Μην πω ξεκινήσαμε πριν από δύο αιώνες. Κάτι αλλάξαμε, κάπως τα επικαιροποίησαμε τα εργαλεία, αλλά είναι τα ίδια εργαλεία. Άρα δεν δουλεύει το σύστημα. Ε, χρειαζόμαστε έναν φορέα ερευνητικό με ευρωπαϊκή προπτική που να είναι ένας πλήρης ευρωπαϊκός ερευνητικός φορέας. Κάποιος αναφέρθηκε σε ένα έμβριο, σε εμβριονικής μορφής φορέα, κάτι που είμαστε εμείς. Είμαστε η αρχή, το βλαστάρι. Πρέπει να αναπτυχθεί ο φορέας. Το ίδιο ισχύει και το Eurojust ερευνητικός φορέας ευρωπαϊκός χρειάζεται και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή εισαγγελία που να έχει το δικαίωμα εκδόσεως εντάλματος και ερευνών. Δεν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αυτό μπορεί να παραμείνει αρμοδιότητα των εθνικών δικαστηρίων. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία να γίνει κάτι τέτοιο, διότι προβλέπεται από τη συνθήκη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη επεξεργάζεται μία πρόταση η οποία θα υποβληθεί επισήμως του χρόνου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υποβληθεί και στο Συμβούλιο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι αυτή η επιτροπή μας, αυτή η επιτροπή, αν με ρωτάτε, κατά την άποψή μου, αν επιτρέπετε, ίσως ανοίξει το δρόμο για κάτι τέτοιο, τουλάχιστον το στο Κοινοβουλίο και αυτό είναι σημαντικότατο. Πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως λοιπόν Μπορούμε να το αναπτύξουμε αυτό. Όλαφ και η Γενική Διεύθυνση Just, θέματα δικαιοσύνη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν επιληφθεί του θέματο και εντό των ε, δύο Γενικών Διευθύνσεων έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά οι μελέτε και εργασίε και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ήδη να το κάνουμε αυτό ατύπω τώρα και να το προτείνουμε στο Κοινοβούλιο. Δεν χρειάζεται να στείλουμε ανώνυμα έγγραφα, διότι ήδη το επεξεργαζόμαστε το θέμα. Το λαθρεμπόριο σιγαρέτων ε, οργανώνεται, είναι οργανωμένο έγκλημα εξορισμού. Ε, απαιτεί αυτή η πράξη επαγγελματική προσέγγιση. Οργάνωση, δεξιότητες, οργανωτικές και επαγγελματικές, εργαλεία, μέσα και οικονομικά μέσα. Σημαντικά, προχωρημένα, πρόκειται περγανωμένου εγκλήματος δεν διαπράττουν κάτι τέτοιο απαραίτητα εγκληματίε που κάνουν άλλα εγκλήματα και μετά κάνουν και λαθρεμπόριο τσιγάρων, παρεμπιπτόντω, για να το πούμε καλύτερα. Τεράστια επιχείρηση. Μεγάλη κλίμακα, τεράστια. Δεν έχω τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν θέλω να πω κάτι από τη, απ' έξω από τη μνήμη μου τώρα. Θα σας στείλω γραπτός. Μπορώ να σας στείλω κάποια στοιχεία που έχουμε αλλά τεράστια κέρδη υπάρχουν. Τα Το κόστος των τσιγάρων, η παραγωγή είναι πολύ χαμηλή. Το κόστος τη παραγωγής είναι πολύ χαμηλό. Μετά όμως ε, οι φόροι αυξάνουν την τιμή. Τα τεράστια... Είναι τεράστια τα κέρδη για εκείνους που κάνουν το λαθρεμπόριο. Η ζημιά λοιπόν για τα οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ενώση οφείλεται σε απώλεια εσόδων. Τελών, εσόδων, των φόρων που εισπράττονται από τα τσιγάρα. Πέρα από τον κίνδυνο που δημιουργείται για την υγεία, διότι πολύ συχνά, αλλά όχι πάντα, το λαθρε... τα τσιγάρα του λαθρεμπορίου είναι πολύ συχνά α, κακέκτυπα. Δεν ξέρει, κα... δεν ξέρει κανείς τι καπνίζει. Δεν, είναι πραγματικά τσιγάρα, πραγματική μάρκα, είναι παραποιημένα προϊόντα. Έχουμε λοιπόν την παραγωγή των ε, σιγαρέτων, παραγωγή καπνού. Άρα είναι επαγγελματίε αυτοί οι άνθρωποι. Και, είναι ειδικευμένε ομάδε του οργανωμένου εγκλήματο που ασχολούνται με αυτό το θέμα, με αυτό το τομέα. Όπου υπάρχει ανάγκη συνεργασία είναι στη μεταφορά, στου τρόπου μεταφορά, στα μέσα μεταφορά. Και εκεί είναι πολύ προχωρημένοι, είναι πολύ οργανωμένοι δεν είναι μόνο υπερεθνική η δραστηριότητά τους, αλλά και διπυρωτική. Ε, τι βλέπουμε λοιπόν, ότι σε κάποιες περιπτώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, ε, τα ίδια μέσα μεταφορών, τα μεταφορικά χρησιμοποιούνται για το εθρεμπόριο τσιγάρων, αλλά ίσως χρησιμοποιηθούν οι ίδιες διαδρομές, η ίδια οργάνωση, ο ίδιος τρόπος για μεταφορά όπλων ή και ατόμων και ανθρώπων. Δεν είναι παράνομο. Αλλά τέλο πάντων, που μπαίνουν παράνομα αυτοί οι άνθρωποι σε μια χώρα. Υπάρχουν λοιπόν συνεργασίες μεταξύ ομάδων. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά το λαθρεμπόριο των σιγαρέτων είναι πολύ επικίνδυνο ζήτημα οικονομικός. Ε, με εξειδικευμένες ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος ασχολούνται με αυτό. Πώς, ορίζουμε το οργανωμένο έγκλημα. Η Όλαφ δεν είναι φορέας καταπολεμήσεως του οργανωμένου εγκλήματος. Εμείς προστατεύουμε τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχουμε, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πραγματικό ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος. Ε, κάναμε αυτή τη μελέτη που προανέφερα το 2009 και 2010, κάναμε τις έρευνές μας λοιπόν και αναλύσαμε τις εκθέσεις μας ένα χρόνο μετά και σας έδωσα κάποια στοιχεία. Παρέθεσα κάποια αριθμητικά στοιχεία στην παρέμβασή μου. Βάση ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος που προέρχεται από δήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης, νομίζω, αν δεν απατώμε, κάτι τέτοιο. Οπότε ακόμα δεν έχουμε καθιερωμένο ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος. Θα έχουμε όμως. τον παρόδο ότι μου έρθει στο μυαλό μια άλλη ανάγκη που έχουμε. Χρειαζόμαστε επίσης κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε σαν Επιτροπή πέρα από τον Ευρωπαϊκό, τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελία χρειαζόμαστε και ποινικό δίκαιο. Ε, ουσιαστικό ποινικό δίκαιο με κοινό ορισμό με κοινού ορισμού για αυτά τα εγκλήματα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποφύγουμε έλλειψη δικαιοδοσίας πώς να το πω, να αποφύγουμε να δώσουμε νομικές δυνατότητες και κενά να τα εκμεταλλευτούν οι εγκληματίες προς όφελός τους λόγω διαφορών ορισμών των ε, εγκλημάτων και δικημάτων ή λόγω έλλειψη ορισμών ή λόγω έλλειψη ποινικοποίηση κάποιων πράξεων σε κάποιε χώρε ή λόγω διαφορών χρονικών ορίων. και στο βαθμό σοβαρότητας κυρώσεων που επιβάλλονται για κάποια εγκλήματα και αδικήματα. Και επειδή θέλουν αποτελέσματα, και είναι επαγγελματίε είναι σοβαροί, διότι κερδίζουν ή χάνουν πολλά χρήματα. Έχουν καλούς δικηγόρους. Προσέχουν, δεν είναι αφελείς. Ακόμα και η μικρότερη διαφορά μπορεί να υπάρχει μεταξύ χωρών και όσον αφορά και το συστικό ποινικό δίκαιο, ε, είναι κάτι που το εκμεταλλεύονται. Λεπτομέρειες, ας πούμε όπως ε, ε χρόνος εδώ στο οποίο πρέπει κάτι να διωχθεί. Πότε παραγράφεται κάτι και εμείς παλεύουμε αυτά τα προβλήματα. Αν θέλουμε να πάμε σε μια δικαιοδοσία και ξέρουμε ότι μετά παραγράφεται σε δύο χρόνια. Γιατί πάμε σε αυτή τη δικαιοδοσία, διότι αποφάσισαν οι εγκληματίες να βάλουν τα χρήματά τους σε αυτή την ε, χώρα για να, να διαφθείρουν κάποιον, Φερρυπίν, κάποιους. Για τα τσιγάρα στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό υπερβαίνει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ακόμα και η προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία αναφέρθηκα και σας ζήτησα μπορεί ενδεχομένω να αποδειχθεί ανεπαρκής γιατί υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα το οργανωμένο έγκλημα που έχει σχέση με το λαθρεμπόριο τσιγάρου. Για τη διαφθορά είναι εργαλείο που χρησιμοποιούν. Παράδειγμα, ακριβώς για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Καμιά φορά χρειάζεσαι να πληρώσει και τίποτα μπαξίσια για να ε, επιταχυνθεί η διαδικασία. Δεν είναι στόχος η διαφθορά, ε, είναι μέσον. Ε, τρόπος διευκόλυνσης των πραγμάτων. Λάδωμα. Ο Περικλής Είναι ένα μικρό σχέδιο με οικονομικούς όρους μεταξύ των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το πιο, τα πιο μικρά. Αλλά είναι ένα από τα δύο προγράμματα που διαχειρίζεται η Όλαφ, όπως γνωρίζετε. Έχουμε αυτό το ταμείο. Δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια, λίγα είναι. Ένα. Εντάξει. Ακριβώς ένα εκατομμύριο, άρα είναι μικρό το πρόγραμμα σε οικονομικούς όρους. Ε, και το διαχειρίζεται όμως η Όλαφ για να αυξηθεί η δυνατότητα των κρατών μελών, όχι μόνο των κρατών μελών όμως, να ανταποκρίνονται, γιατί είναι πολύ ευρύτερο το θέμα και πάλι υπερβαίνει τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την παραχάραξη του ευρώ, ε, ιδιαίτερα των ε, νομισμάτων ε, και των τραπεζογραμματίων. Είναι λίγα χρήματα, αλλά πιάνουν τόπο. Γιατί δεν χρειαζόμαστε πολλά λεφτά σε αυτή την προσπάθεια. Εκπαιδεύουμε υπαλλήλου ε, και της Ένωσης και εξοκοινοτικούς, ιδιαίτερα σε χώρες που είναι πιο επικίνδυνη αυτή η ε, παραχάραξη του ευρώ, για να δημιουργήσουμε και ένα διεθνές δίκτυο ε, διεκτικών αρχών με ιδιαίτερη δίκευση σε αυτό το θέμα. Και λειτουργεί καλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται εδώ πάρα πολλά χρήματα. Νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Όλαφ είναι πολύ γνωστή μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. <laughs> Εντό και εκτό της ενώσεω για τη δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και Διευθυντά. Έχουμε τελευταίο αίτημα για μιλία, ερώτηση-απάντηση. Η κυρία Λάτφορντ έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο Διευθυντής. Θέλω να τον πιέσω λίγο παραπάνω. Ε, μπορεί να χρειάζεται βεβαίως εναρμόνιση ε, κάποιων ε, στοιχείων του ποινικού δικαίου στην Ένωση για να ε, μπορούμε ε, να μην αφήνουμε τους μεγαλογκληματίες να εκμεταλλεύονται τα κενά και τα ελλείμματα. Υπάρχουν ορισμένοι κόμματα και ομάδες που λένε απαράδεκτη απώλεια κυριαρχίας αυτό το πράγμα. Όχι, αξίζει τον κόπο ε, να πιάνουμε τους εγκληματίες. Και αυτοί που αντιτίθενται σε αυτή την εναρμόνιση νομίζω δεν μπορούν να ισχυρίζονται ότι είναι υπέρ της τάξης και του νόμου. Δεν θα τους κατονομάσω, αλλά καταλαβαίνουν ήδη ποιοι είναι. Το άλλο θέμα, όμως του Ευρωπαίου εισαγγελέα, νομίζω ότι είναι λιγότερο πιστικό για μένα. Μιλήσατε για μια εισαγγελία που να έχει και διοκτικές αρμοδιότητες. Αυτό όμως θα εξαρτάται ακόμα από τη συνεργασία ε, εθνικών διεκτικών αρχών αστυνομία και εισαγγελία. Εγώ δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτό το σύστημα ε, θα λειτουργούσε εφόσον δεν λειτουργεί Eurojust γιατί και εκεί χρειάζεται συνεργασία αστυνομία με τη δικαιοσύνη και γνωρίζουμε και με τους εισαγγελείς προκειμένου ότι οι αρχές των κρατών μελών δεν δείχνουν αρκετή προθυμία να το κάνουν. Όπως επίσης δεν δείχνουν αρκετή προθυμία ε, να δίνουν στη Europol αρκετά στοιχεία κλπ. Λοιπόν, πώς θα μπορούσε μια ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ε, εξακολουθεί να εξαρτάται από τη συνεργασία των εθνικών κρατών, πώς αρχών, συγγνώμη, θα λειτουργεί καλύτερα από την ε, Eurojust. Δεν είναι τόσο ιδεολογική η αντίρρησή μου, είναι πάρα πολύ πρακτική φύσεως. Θα λυθούν όμως τα προβλήματα, πανάκια, είναι Ευρωπαίος εισαγγελέα, Πώς θα λειτουργήσει και γιατί θα λειτουργήσει καλύτερα από τη Eurojust που δεν λειτουργεί αρκετά καλά. Uh, I, I see the point. Εντάξει, το καταλαβαίνω το ερώτημά σας, λέει ο κ. Είναι κρίμα που πρέπει να το συζητήσουμε μόνο σε μερικά λεπτά, διότι πίσω από αυτό, πίσω από το ερώτημά σας και πίσω από την απάντησή μου, κρύβεται μεγάλος προβληματισμό και δουλειά. Τέλο πάντων, πρώτα απ' όλα. Πρώτον, νομίζω ότι θα πρέπει να μετακινηθούμε από προσέγγιση συνεργασίας, δηλαδή Eurojust, που συνεπάγεται εθνική επεξεργασία του θέματος και απλώς συνεργασία τα εθνικών φορέων, αλλά γενικότερα η κίνηση γίνεται στο εθνικό επίπεδο. Εθνική προσέγγιση συνεπάγεται συνεργασία. Να πάμε από τη συνεργασία σε αυτό που θα έλεγα εγώ ολοκληρωμένη προσέγγιση, αν το προτιμάτε. Πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Κάτι που χρειάζεται και πολύ μάλιστα. Σαν σύλληψη, σαν έννοια είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε τώρα. Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Συγγελίας που έχει εξουσίες ερευνητικές και δικαστικές εντολές, δικαιώματα, δικαιοδοσία. Έρευνα, δίωξη. Ε, δεν το προανέφερα γιατί εστιαζόμουν στο τέλος του θέματος, αλλά χρειάζεται συνεργασία με εθνικούς ερευνητικούς φορείς, δηλαδή αστυνομικέ υπηρεσίες και εθνικές εισαγγελίε. Και στο μοντέλο που αναπτύσσουμε στις συζητήσεις μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχουν προχωρήσει συζητήσει. Φανταζόμαστε αυτή την υπηρεσία αρκετά μικρή, ω μέγεθο μικρή υπηρεσία, ευρωπαϊκή υπηρεσία που θα βασίζεται επί δικτύου, δικτύου ε, εθνικών διοκτικών φορέων, εθνικών εισαγγελιών, συγγνώμη. Οπότε έχουμε ακόμα εθνική προσέγγιση, εθ, δικτυωμένοι οι φορείς και δικτύωση με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Εν κατακλείδη, περί αυτού πρόκειται, επεξεργαζόμαστε λεπτομέρειες. Δεν έχει ως ευθύνε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέα και οι δικαστικέ αρχές των κρατών μελών ε, έχουν απεκτηθεί των ευθυνών του. Αντιθέτω θα ενταχθούν σε ένα δίκτυο, θα δικτυωθούν μεταξύ τους μαζί με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Οπότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Υπηρεσία απαρτίζεται από μια μικρή υπηρεσία, θα βρίσκεται κάπου στην Ευρώπη, δεν θα πω ποτέ πού, αλλιώς θα δεχτώ πειρά, θα κινδυνεύσω. Κάπου στην Ευρώπη θα εδρεύει η κεντρική υπηρεσία και θα απαρτίζεται από εθνικές υπηρεσίες που οργανώνονται στα πλαίσια εθνικού δικαίου ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αυτό πρέπει να είναι το, το, το μοντέλο που προβλέπω, που διαβλέπω. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, πόρο απέχουμε από μία απόφαση, αλλά αυτή είναι η ιδέα την οποία επεξεργαζόμαστε. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας, κύριε Διευθυντά, αλλά κυρίω για αυτά που μα είπατε και για σημαντικά στοιχεία που μα αναφέρατε, κυρίω και για την εντολή τη Επιτροπή και γιατί υπογραμμίσατε την ανάγκη που υπάρχει κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στη διάθεσή της ε, μια σοβαρή νομοθεσία καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος τύπου μαφίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Εάν οργανώνεται το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να οργανωθούν και οι θεσμοί για την αντιμετώπιση του. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα περνούμε στην επόμενη ε, παρουσίαση είναι κάποιος ε, που εργάζεται επί τόπου, είναι εκτεθειμένος κάθε μέρα και μαζί με την πείρα του ε, θα μας πει τι συμβαίνει με το οργανωμένο έγκλημα και τη μαφία. Αλφόνσο Νταλφόνσο είναι διευθυντής ε, της Ιταλικής Αρχής κατά της μαφίας και της διοκτικής αρχής Interforce που ασχολείται με καταπολέμηση της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Καλό το Διευθυντή να μας κάνει μια σύντομη παρουσίαση, όχι μόνο σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των Ιταλικών μαφιόζικων οργανώσεων, αλλά κυρίως των εγκληματικών οργανώσεων ε, που δρούν ε, στην Ιταλική επικράτεια και ε, πώς εκτείνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς μπορούν να ε, παταχθούν και να εκριζωθούν. Ε, και το ίδιο θα ισχύσει με την προηγούμενη τοποθέτηση. Θα μας κάνει τη εισαγωγή ο Διευθυντής, μετά οι βουλευτές, μετά θα ξαναπαντήσει και χρειαστεί δεύτερος γύρος ερωτήσεων. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας παρουσιάσω γενικά ε, τα θέματα ε, και μερικά στοιχεία για να καταλάβουμε καλύτερα κάποιες βασικές αρχές. Ποιος είναι ο στόχος να υπογραμμίσουμε ότι ε, σήμερα μπορεί να διαπιστώνουμε κάποιες πρόοδους στην καταπολέμηση αλλά προχωρούν και οι εργανώσεις αυτές. Υπάρχει μια σιωπηρή διείσδυση ε, και ε, των οργανώσεων αυτών είναι πολύ καλά οργανωμένες. Αυτό το ε, έδειξαν και οι έρευνες που έκανε η υπηρεσία μας εντάσσονται σε πολύ διαφορετικές κοινωνικές πραγματικότητες και εδαφικές. Δεν χρειάζεται να ελέγχουν στρατιωτικά, ας πούμε, ένα ε, χώρο, αλλά με διείσδυση ε, επιτόπου και τους αποφέρει αυτό πολλά έσοδα. Ε, μιμούνται τις νόμιμες δραστηριότητες, τις αντιγράφουν και γι' αυτό μένουν ε, χωρίς να αποκαλύπτονται. Αυτό είναι και η κόζα νόστρα ε, που είναι σαν ένα χταπόδι που απλώνει τα πλοκάμια του παντού. Έτσι οργανώνεται η εγκληματικότητα που σε μεγάλο βαθμό είναι αόρατη ή σιωπηρή. Γνωρίζετε και δεν χωρά καμία αμφιβολία στην Ιταλία ιστορικά έχουμε μαφιόζικες οργανώσεις που είναι ε, καλά ριζωμένες σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, στη Σικελία αλλά και στην Καλαβρία, στην Καμπανία και στην Απουλία. Κοζανόστρα ονομάζεται μαφία ανάλογα. Ε, η Τζάγκετα στην Καλαβρία, η Σάντα Κορώνα Ουνιτά ε, στην Απουλία και η Καμόρα στην Νάπολη. Αυτή όμως η εδαφική του συγκρότηση και οι ρίζες τους συνοδεύονται και από μια ευρύτερη παρουσία που είναι πολύ λιγότερο οργανωμένη σε άλλες περιφέρειες. Ε, υπάρχει και ε, αλλαγή ε, και εξέλιξη σε άλλες περιφέρειες της Ιταλίας που είναι το Πεδεμόντιο, η Λομβαρδία, η Λιγουρία στο παρελθόν, η Εμιλία Ρωμάνια που δεν υπήρχαν αλλά σήμερα έχουν διεισδύσει μέχρι και αυτές τις περιφέρειες. τα εθνικά αντισώματα που κανονικά θα μας επέτρεπαν να καταπολεμούμε αυτή την αρρώστια ήταν νομοθετικού χαρακτήρα για να μπορούμε καλύτερα να ξέρουμε τι χρειάζεται να υιοθετήσουμε ε, για να καταπολεμήσουμε αυτό το οργανωμένο έγκλημα νέου είδους. Τελικά θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο πώς να το πω, στη διάδοση εγκληματικής είναι δύσκολο να ανοιχνευτεί γιατί ε, είναι εγκιστρωμένο στην τοπική οικονομία και έχει άμεση επίπτωση και στην ασφάλεια και γενικότερα η ανάλυση γίνεται βάση ε, της ζημίας που υφίσταται η οικονομία που δεν είναι ο καλύτερος τρόπος ανάλυσης αυτός. Λοιπόν, και έχουμε περάσει από ε, στιγμές ε, πάρα πολύ ε, δύσκολες. Περάσαμε από το επιχειρησιακό επίπεδο σε ένα επίπεδο ε, ένταξη στην νόμιμη οικονομία. Αυτή η διάδοση και η διάχυση στην εθνική επικράτεια είναι ένα από τα περάσματα. Ε, γι' αυτό εγώ λέω σήμερα ότι ο αντίκτυπος αυτού του είδους της εγκληματικότητας δεν πρέπει να υποτιμάται διότι είναι κάτι που ήδη λειτουργεί σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ε, ε Ένωσης. Γίνονται διάφορες έρευνες αυτά τα χρόνια. Ε, ε βλέπουμε διάφορα διάφορες ε, αξιολογίες που γίνονται στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, ε, στα Βαλκάνια, όπου υπήρξαν εκεί δραστηριότητες που μεταφέρθηκαν από την Ιταλία σε αυτές τις χώρες με τα ίδια χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, του Ιταλικού οργανωμένου εγκλήματος. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, πιστεύω, πώς να το πω, ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή, πιο εστιασμένη προσοχή, στις συνέπειες που έχει το οργανωμένο έγκλημα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ξεκινήσω από την Τραγκέτα, τη διεθνή παρουσία της Τραγκέτα. Είναι πάντα πιο παρούσα στην υπηρετική Ευρώπη, στο κοινωνικονομικό επίπεδο. Οι συλλήψεις που έγιναν το 2009 στην Ολλανδία, κάπου κοντά στο Άμστερνταμ, σε σχέση με τον Τζοβάνι Στράντζο και τον Φραντζέσκο Ρωμαίο, τον κουνιάδο του, αποδεικνύουν για ακόμη φορά ότι η Ολλανδία είναι ένας τόπος που ενδιαφέρει ε, μια ομάδα και εκεί κινούνται οι πιο επικίνδυνοι ε, και συμμετείχαν αυτά τα μέλη ε, στην σφαγή στο Ντούισμπουργκ. Στη Γερμανία πιστεύουν ότι υπάρχουν ε, δίκτυα της Ντράγκετα που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 70 και έχουν βγάλει ρίζες, έχουν πια στη Γερμανία. Η συνεργασία με την Bundeskriminal, την υπηρεσία την εγκληματολογική της Γερμανίας, δείχνει ότι χρειάζεται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της Ιταλικής Ομάδας Εργασίας και τις υπηρεσίες που λειτουργεί στη Γερμανία που δημιουργούν την Task Force που δημιουργήθηκε μετά τα γεγονότα του Duisburg του 2007 που οδήγησαν στην ε, περίφημη φάιντα τη Σαν Λούκα. Είναι ένα χωριουδάκι το Σαν Λούκα στη, στην Καλαβρία, στο Ρέτζο Καλά. Ε, παρήγαγε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις τύπου μαφίας. Άλλο σημαντικό επεισόδιο είναι η σύλληψη στην Ισπανία ενός Ιταλού ε, που ε, τον έψαχναν σε όλη την ε, διεθνώς για το ελευθερμπόριο ναρκωτικών. Σχετιζόταν με τράγκετα και στην Ισπανία είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο κίνηση κοκαίνη κοκαίνης που μέσω υβηρική, από Ιβυρική Χεσόνησο πήγαινε στην Ιταλία. Λοιπόν, δεν πρέπει να λησμονούμε λοιπόν ότι η προτιμησιακή διαδρομή κυρίως της Ντράγκετα είναι η μεταφορά ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική προς Ισπανία και μετά πηγαίνουν στην Ιταλία τα ναρκωτικά. Αλλά και η Καμόρα έχει κλάδους, παρακλάδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τις οργανώσεις τύπου Καμόρας το λαθρεμπόριο ναρκωτικών προς την Ιταλία από τις χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης είναι το πιο επικερδές λαθρεμπόριο. Λοιπόν, και δείχνει ότι υπάρχει προτίμηση Ισπανίας για τη διέλευση. Η παρουσία της Καμόρας στην Ισπανία ε, έχει, είναι πολύ σημαντική. Η Κώστα Τελσόλ, η Κώστα Μπράβα ε, έχουν οργανώσεις τύπου Καμόρας με αρνητικότατες συνέπειες για την τόπια οικονομία και μέσω επενδύσεων στα ακίνητα κινούνται κάποιες ομάδες χρησιμοποιώντας κεφάλαια από παράνομες πηγές. Και στην Ολλανδία υπάρχουν κλάδοι της Καμόρα, στη Ρουμανία και ούτω καθεξής. Στη Γερμανία υπάρχουν και δραστηριότητα της Καμόρα στο εμπόριο προϊόντων α, παραποιημένων που κατασκευάζεται βασικά στην Κίνα. Σε αυτό το πλαίσιο, στο Αμβούργο, Μόναχο και στο Ντόρμοντ ε, βρίσκονται, αλλά υπάρχουν και διάφορες ομάδες που σχετίζονται με ε, ομάδες της ε, Νάπολης, στην Κολονία, στην Φραγκφούρτη και στο Βερολίνο και στην Πολωνία. Υπάρχουν. Αυτή είναι μια πανοραμική εικόνα λοιπόν που μας δείχνει να καταλάβουμε ότι το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Είναι πολύ εξωσημείωτες, μεγάλες, ε, φοβερές οργανώσεις που έχουν δυνατότητα δίσδυσης. Όχι μόνο στη χώρα, σε μια επικράτεια, αλλά στο κοινωνικονομικό, στον κοινωνικονομικό ιστό μιας χώρας. Και αυτή την περίοδο της μεγάλης οικονομικής και χρηματοστικής κρίσης πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί διότι είναι ακόμα πιο ε, επικίνδυνο αυτό το εγκληματικό σύστημα που τίνει να υπονομεύει τα θεμέλια της νόμιμης οικονομίας. Και στην Ιταλία υπήρξε υποτίμηση του φαινομένου της μαφίας. Όμως σήμερα ε, έχουμε τις απαρχές του συστήματος καταστολής του φαινομένου. Έχουμε νομοθεσία που θέλει να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Στα πλαίσια του ποινικού κώδικα έχουμε το άρθρο 416α που αφορά τις ενώσεις τύπου μαφίας και ξένες ομάδες τύπου μαφίας. Και έχουμε δώσει ορισμό της ποινική οργάνωσης και περιγράφονται και οι μηχανισμοί λειτουργίας. Και ξεπεράσαμε τα όρια του, του, του, του άρθρου του ποινικού κώδικα του 416, δηλαδή που αφορούσε τις ενώσεις ε, για διάπραξη αδικημάτων. θα πρέπει να διαπιστώνεται τη διάπραξη των αδικημάτων και ότι οργανώνονται σε ομάδα για να διαπράξουν συγκεκριμένε πράξεις. Κίνδυνο για δημόσια ασφάλεια. Λοιπόν, ευδημιουργούνταν παλιά κενά από τους ορισμούς και τώρα προσπαθούμε να τα καλύψουμε και να αντιμετωπίσουμε τις πιο σύγχρονες εκδηλώσεις του, των μαφιόζικων οργανώσεων. Λοιπόν, αφορά, λοιπόν, οι αλλαγέ όσον αφορά το άρθρο 416 του ποινικού κώδικα. Λοιπόν, καθορίζει τη διαφορά, διότι η οργάνωση τύπου μαφίας υπήρχε και πριν την διάπραξη συγκεκριμένων αδικημάτων. Ένα άλλο εργαλείο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πετόπιση της ε, εγκληματικότητας αυτής είναι ο εντοπισμός των προληπτικών μέτρων σε προσωπικό επίπεδο και κλήρωση όσον αφορά τα στοιχεία τα περιουσιακά που συνοδεύουν την ποινική δίωξη και, και βασίζεται η υλοποίηση του μέτρου αυτού στην ε, λογική υπόνοια, αν θέλετε, τη βάσιμη υπόνοια, αντί της ύπαρξης απόδειξης, επί του οποίου στοιχείου βασιζόταν το ποινικό δίκαιο. Πρόκειται περί ε, δικαστικής προσέγγισης αφορά την κατάσχεση, που εξασφαλίζει και την σωστή προστασία των τρίτων μερών που καλή την πίστη είχαν σχετιστεί με αυτούς, χωρίς να το ξέρουν. Λοιπόν, όσον αφορά την ποινική δίωξη και την φυλάκιση, το άρθρο 41α αφορά την ε, κάθερξη. Λοιπόν, για να ξεκινήσει αυτή η ποινική δίωξη, χρειάζονται να χρησιμοποιούν όλα τα διάφορα μέσα που είναι στη διάθεση των ε, αρμοδίων αρχών και των δικαστικών αρχών. Πιστεύουμε λοιπόν γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο πρέπει να πω ότι πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του φαινομένου του οργανωμένου εγκλήματος δημιουργηθεί μια μονάδα ανάλυσης δίπλα στη Europol μαζί με τις ειδικευμένες άλλες αρχές της Ιταλικές θα μπορούσε να βοηθήσει και να υποστηρίξει στην υλοποίηση της πρωτοβουλία χρησιμοποιώντα όλη την τεχνογνωσία και την εμπειρία που υπάρχει όσον αφορά τη μαφία. Μπορεί να δημιουργηθεί εντός των ευρωπαϊκών δομών, στα πλαίσια της Europol, ένα ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρησιακό καταπολέμησης των οργανώσεων αυτών τύπου μαφίας, που θα επιτρέπει καλύτερη εφαρμογή και ένταξη της ερευνητικής πτυχής των ερευνητικών διαδικασιών. Αυτά και περιμένω ερωτήσεις. Ε, Οι συντονιστές έχουν το λόγο. Ματιό. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά για την εξαιρετική σας παρουσίαση και σε εθνικό επίπεδο και τις προτάσεις σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στις προτάσεις που κάνατε για τη δημιουργία μιας ε, ενότητας κατά του εγκλήματος στην Ευρωπόλ. Είναι μια πρόταση που ειλικρινά θα μπορούσε να έχει γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια ερώτηση. Από πότε δραπιστώσατε την επέκταση της οργανωμένου κλίματος στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και για σας ποια είναι η άποψή σας η επέκταση αυτής της εγκληματικότητας είναι γιατί χρειάζεται εξουσία, δύναμη, η μαφία ή ανάγκη χρημάτων. Είναι δηλαδή η οικονομική διάσταση ή η εξουσία, η διάσταση εξουσίας. Κάτι που αισθάνονται σαν ανάγκη ενδεχομένω συνωνεί. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω αν έχετε δει κάποια εξέλιξη από τον τελευταίο πόλεμο ή έχει να κάνει μια, την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ε, τελευταία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Φαγιόν για το S&D. Κυρία Φαγιόν. Ευχαριστούμε και το Διευθυντή για τις διευκρινήσεις που μας ε, έκανε. Πάρα πολύ καλές διευκρινήσεις και εξηγήσει όσον αφορά τις ε, οργανώσεις αυτές τύπου μαφίας και τη δραστηριότητά του στην Ευρώπη και στο διεθνέ προσκήνιο. Αναφερθήκατε στην Πολωνία, στη Γερμανία, στα Δυτικά Βαλκάνια όσον αφορά τη δραστηριότητα της μαφίας. Ποια είναι η συνεργασία των ερευνητικών αρχών ε, με, και μαζί σας οι αρχές των χωρών που είναι καθοδόν προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστυνομικέ αρχές ε, ίσως δεν είναι ακόμα τόσο αποτελεσματικές οι χώρε όσο θα έπρεπε. Ποια προβλήματα δια, βλέπετε όσον αφορά την, ε, τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και ενδεχόμενη ένταξή τους. Τον επόμενο μήνα θα πάμε στη Σερβία. Αντιπροσωπεία θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τους αρμόδιους φορείς της Σερβίας. Λοιπόν, από πλευρά σας θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια σχόλια όσον αφορά την κατάσταση ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία δημιουργίας Ευρωπαϊκού Δικτύου για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Θα με ενδιαφέρει να γνωρίζω ε, ποια είναι η θέση σας βλεβάνοντας υπόψη και την εντολή που έχει δοθεί στην Επιτροπή ΚΡΙΜ. Χρειαζόμαστε πράγματι μία εντολή, να υπάρξει μία εντολή για τον Ευρωπαίο Σαγγελέα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νιούτον Τόν έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι, με ψάχνετε. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Εγώ που δεν είμαι Ιταλός, όπως περισσότεροι, σε αντίθεση μάλλον με τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής, ομολογώ με μεγάλη μου ντροπή. Ε, θέλω να σας ρωτήσω πώς λειτουργούν αυτά. Ε, σε οικογενειακή βάση Δηλαδή θα στείλω στο Μιλάνο τον αδελφό μου ή τον ξάδελφό μου στην Κώστα Μπράβα. Ποιος είναι ο μηχανισμός εμπιστοσύνης, εχημήθειας ή προσλαμβάνουν αλλοδαπούς. Και στη συνέχεια, ποια είναι η σχέση μεταξύ της μαφία, της καμόρα, της δράγκετα και το ε, ε, λοιπόν, είναι εχθροί, θανάσιμοι εχθροί, συνεργάζονται, πώς λειτουργούν οι οργανώσεις για Πολύ σύντομα. Θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με την κυρία Φαγιόν. Αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι αυτό που είπατε για την αναδυόμενη οργανωμένη κλιματικότητα από τη Δυτικά Βαλκάνια. Είναι μια επικράτεια εκτός της Ένωσης και θα ήθελα να μας πείτε λίγο περισσότερα για τη συνεργασία, για την έλλειψη συνεργασίας και είναι σημαντικό γιατί θα πάμε και στη Σερβία και πρέπει να προετοιμάσουμε καλά αυτή την επίσκεψη. Ε, και τώρα για την Κουε, ο κ. Σαντεργκάντ έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Δευθυντή για την παρουσίασή του. Έχω αντίστοιχη ερώτηση. Για τις διασυνδέσεις αυτές Ε, η βεντέτα του Σαν Λούκα, από ό,τι κατάλαβα, ξεκίνησε εκεί και μετά επεκτάθηκε. Αλλά υποθέτω ότι δεν σκοτώνονται 16 χρόνια μετά για αυτό το πράγμα οι άνθρωποι. Γιατί διαδόθηκε και πώς διαδόθηκε. Και αυτό αφορά ε, και άλλους κατοίκους της χώρας ή μόνο τους Ιταλούς και την Ιταλική μαφία. Ε, και έχω και μια ερώτηση, καλύτερα ένα δίλημα. Γιατί το θεωρώ λίγο παράδοξο. Μια χώρα η οποία έχει την περισσότερη νομοθεσία κατά της μαφίας ε, και τους περισσότερους περιορισμούς και τις περισσότερες διώξεις και, μας περιπτώσει, την περισσότερη εμπειρία και αστυνομικούς, είναι η χώρα όπου είναι η ισχυρότερη μαφία. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο. Και σε σχέση με αυτό, ε, ε μπορεί να μας πει ο Διευθυντής κάτι ε, για τη σύνδεση, η διασύνδεση των μαφιόζικων δραστηριοτήτων με την πολιτική. <laughs> δηλαδή, σε ποιο βαθμό η μαφία μπορεί να επηρεάσει το πολιτικό σύστημα και το νομικό σύστημα. Ε, και ε, τη δικαστική ατζέντα, τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Μπορεί η μαφία να επαγορεύει νόμους, ας πούμε. Μπορεί να επαγορεύει ε, τις δικαστικές αποφάσεις. Ε, πώς το εκτιμάτε αυτό. Μάκιντάρ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Κυρία Μακιντάρ. Ε, είδα ότι κατέφτασε δικός μας ε, συντονιστής, αν θέλει να μιλήσει, ε, να του αφήσω το λόγο. Δεν θα μιλήσω εγώ. Όχι. Καλά. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Και εγώ μιλώ ως μη Ιταλίδα. Είμαι μέλο τη Επιτροπή ε, Μειοψηφία, αλλά περνάω όλε μου τι διακοπέ στην Ιταλία και αισθάνομαι έτσι κάποια συγγένεια και κάποια συμπάθεια. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Χρειάζεται ειδική μονάδα στη Europol για την καταπολέμηση της μαφίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Πώς ε, το αξιολογείτε αυτό. Θα δώσει προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση του εγκλήματος. Τι μπορούμε εμείς να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πώς λειτουργεί καλύτερα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αντίθεση με το εθνικό. Eh, e. Και τώρα για το ΕΛΚ. Για ένα λεπτό, δύο Μέρα, Κύριος Μέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν μιλώ εξ ονόματος του ΕΛΚ, η Βερονίκ Ματιού μιλάει εξ ονόματος του ΕΛ και εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Θα ήθελα να πω στον κύριο Αλφόνσο ότι μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίασή του. Κατανοώ πάρα πολύ καλά αυτά που λέτε και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε και τα μηνύματα που στέλνετε. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας σε τούτη εδώ την Επιτροπή. Ε, πολύ ωραία τα λόγια σας και μου αρέσουν πολύ γιατί θα καταλάβει και η Επιτροπή την πρόταση που έκανα εγώ αρχικά. Πιστεύω κύριε Αλφόνσο ότι το έγκλημα έχει υποστεί σημαντική εξέλιξη και οι μαφίες οι ίδιες. Και εσείς γνωρίζετε πολύ καλά όπως και εγώ ότι πρώτον πρώτα μπήκανε στο τζόγο μετά, στο τζόγο, μετά πήγανε στο αλκοόλ και τώρα έχουν φτάσει στα ναρκωτικά και τι γίνεται στις χώρες προέλευσης και ε, διέλευσης ε, ή μέχρι τις χώρες ε, αποστολής. Δηλαδή είναι μια λυσίδα ολόκληρη. Παραγωγή, διαμετακόμιση και τελικός προορισμός. Και η χώρα σας, η Ιταλία και η δική μου Ισπανία είναι και χώρες διαμετακόμισης και χώρες προορισμού. Δηλαδή φέρνουν και το προϊόν εγκλήματος ε, στις χώρες αυτές και το διαδίδουν και το διακινούν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα ήθελα λοιπόν να έρθουν εμπειρογνώμονες ε, των χωρών προέλευσης, αλλά και να τις επισκεφτούμε αυτές τις χώρες. ήθελα ε, να ρωτήσω και αυτό που ρώτησε η κυρία Μάκιντάιρ. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μια αντία σαν την DEA των Ηνωμένων Πολιτειών στο εσωτερικό της Europol. Δεν νομίζω, γιατί τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που γνωρίζουν καλύτερα και περισσότερα τους τρόπους δίωξης και πάταξης της μαφίας. Και επίσης η Ευρωπόλ έχει περιορισμένες ε, ε, δυνατότητες, τελειώνω πρόεδρε, και εξουσίες. Είναι καλή ιδέα πλην ανεφάρμοστη διότι γνωρίζετε ότι τα κράτη-μέλη είναι πολύ καλά στο να ε, κρατούν τις προφορίες τους και να μην τις μοιράζονται με άλλους όταν πρόκειται για διώξεις. Ενώ για την καταστολή δίνουν πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ ε, που ήρθατε και ήθελα να κάνω μόνο αυτό το σχόλιο. Και τώρα τελευταία παρέμβαση. Ο κ. Σωσέτα έχει το λόγο συντομότατα κάποιες ερωτήσεις έθεσαν. Λοιπόν, ε, μπορείτε να απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις που πολύ συχνά τίθενται από διάφορους συναδέλφους. Ε, συνδέθηκα με, την ιστοσελίδα ε, όπου γίνεται μια καταγγελία στο παρέλβο Λοιπόν, στη, ο, ο Μπόσλαν Κατόρε είχε δραστηριοποιηθεί στο Λονδίνο. Η Αγγλία αρνήθηκε σε ένα πιο επικίνδυνο μαφιόζου, επικεφαλή τη μαφία τη οικογένεια στην Τραμπία, που, κοντά από το Παλέρμο, να δώσει την έκδοση στην Ιταλία. Παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί για πολύ με, πάρα πολλά δικήματα. Μα εμείς με την κυρία Μπορσελίνο και λοιπά επανειλημμένα είχαμε θέσει αυτή την ανάγκη που υπάρχει. Κατά κάποιο τρόπο το αδίκημα τύπου μαφίας να περιγράφεται σαφέστερα. Διότι στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης η έκδοση δεν μπορεί να απορριφθεί για ε, αδικήματα. Δεν μπορεί τα κράτη-μέλη είναι μια ένωση εγκληματική μαφία. Θα πρέπει να αναγνωρίζετε ότι υπάρχει μια οργάνωση εγκληματική που έχει τέτοιες... Όταν ε, κάποιος ανήκει σε μια οργάνωση που έχει αυτούς σκοπούς, πρέπει να γίνεται η έκδοση. Δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά την νομοθεσία των κρατών μελών. Πρέπει να διευκρινιστούν οι νομοθεσίες, να είναι ξεκάθαρες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, πολύ συχνά όσον αφορά την ανάλυση αυτών των ομάδων τύπου μαφίας, όχι μόνο τύπου Ιταλικού, ο Ζαν Φρανσουά Γκεϊρό θα μας πει περισσότερα για αυτές τις ομάδες, γιατί έχει μελετήσει το πρόβλημα. Στις ερωτήσεις ε, γίνεται πάντα αναφορά παράμεσα στηριότητα, στα ναρκωτικά κλπ. Όμως πολύ λίγο αναφέρεται το ότι τα εγκληματικά συστήματα και κυρίως τα συστήματα, οι ομάδες που εμπνέονται από τη μαφία είναι ένα σύνολο εντός του οποίου υπάρχει το έγκλημα, η πολιτική και η οικονομία. Δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε μόνο ότι αυτοί που ασχολούνται, ότι ασχολούνταν μόνο με τα αλκοόλ παλιά, ασχολούνται με την, με την κερδοσκοπία, ε, μάλιστα ασχολούνταν με, την, με τα οικονομικά, με τα όπλα κλπ. Εδώ και έναν αιώνα είχαν ξεκινήσει αυτές τις δραστηριότητε. Ε, κύριε Φιντάκη, και οι ερωτήσεις όλες ε, συγκλίνουν επί μιας ανάγκης που υπάρχει. Εγώ απευθύνω έκκληση σε όλους. Έχουμε ήδη 30 λεπτά καθυστέρηση σας. παρακαλώ πάρα πολύ να συγκρατηθείτε στον αφορά το χρόνο που μιλάτε. Λοιπόν, δράτω με τις ευκαιρίες να σας υποβάλω ένα συντομότερο ερώτημα. Ε, πολύ συχνά ζητείτε κάτι υπογράμμισε και ο κ. Σκοτσέτα μας ζητείτε πολύ συχνά τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει σαν βασικό τη στόχο να διευκολύνει την εναρμόνιση των διαφόρων δικαστικών συστημάτων εντός της Ένωσής μας, ούτως ώστε να μπορούμε μετά να πετύχουμε με τον απλούστερο τρόπο και κυρίως προς κοινών όφελος των 500 εκατομμυρίων πολιτών που εκπροσωπούμε, να πετύχουμε, λέγω, ένα νομοθετικό κείμενο, να έχουμε ένα νομοθετικό κείμενο που για μια φορά να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Πιστεύετε ότι είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του οργανωμένου σε κρίζωση των μαφιών, εάν κάθε χώρα ε, έχει δική της ένομη τάξη δικό της νόμο, δικό της κείμενο που διαφέρουν μεταξύ τους ε, σε σχέση με αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Απάντηση. Ζητώ συγγνώμη. Εάν θα είμαι εξαιρετικά συνοπτικός, αλλά ο διαθέσιμος χρόνος είναι ελάχιστος. Το να δώσω απαντήσεις πιο εξαντλητικές επί του πρώτου θέματος για να μπορέσω να εξηγήσω τι είναι οργανωμένο έγκλημα τύπου μαφίας και ε, ποια είναι η δυνατότητα να αναπτυχθεί και σε άλλες χώρες και όχι μόνο ευρωπαϊκές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και μετά ενδεχόμενα διορθωτικά μέτρα που σαν Ευρώπη μπορούμε να εθετήσουμε. Πάνω σε αυτό θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ. Η ιστορία κυριαρχεί στη ζωή μας, ε, ελέγχει τη ζωή μας. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η Σικελία εξήγαγε αναπαράγοντας τη δομή της από τη συγκελία της, της δομή της στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή του είδους η εγκληματικότητα είναι μια εγκληματικότητα που δρά πάντα επί δύο μετόπων. Ριζώνει στην επικράτεια, οπότε βρίσκει κοινωνική συνένεση και ταυτόχρονα εντάσσεται στην οικονομία, την νόμιμη οικονομία ιστορικός πώς υπάρχουν ομάδες, για να μιλήσουμε και για την Τράγκετα, που προσανατολίστηκαν παρομοίως και πήγαν στον Καναδά, πήγαν με τον ίδιο τρόπο στην Αυστραλία. Οπότε ιστορικά ήδη έχουμε αυτά τα περάσματα. Και πρέπει να πω ότι η Ιταλική νομοθεσία που αναπτύχθηκε και δεσπίστηκε τα τελευταία χρόνια ήταν πάντα καρπός μιας νομοθεσίας που ορίμασε ε, λόγω κατεπίγους ανάγκες. Κάποιοι νόμοι, ο πιο σημαντικός νόμος ε, για τις ένωσεις ε, των ομάδων αυτών κλιματικών που έδωσε τη δυνατότητα στην, ε, στη χώρα τη δυνατότητα να κατασχέσει την, τα, τους σπόρους που είναι αποτέλεσμα εγκληματικών πράξεων της μαφίας. Δηλαδή, χρειάζεται πραγματική δράση για να αντιταχθούμε σε αυτό το έγκλημα που δεν πρέπει να υποτιμάται, επαναλαμβάνω, διότι μπαίνει στα ίδια τα γάγκλια της ε, κοινωνίας και διαφθείρει ε, τη διοίκηση και μπορεί να έχει σχέσεις και με την πολιτική. Είχαμε μια, μια σειρά ε, δικαστικών υποθέσεων όπου είδαμε ότι οι πολιτικοί σε διάφορα επίπεδα είχαν εμπλακεί σε αυτούς τους μαφιόζικους μηχανισμούς. Γι' αυτό τώρα πια έχουν ήδη ε, γίνει δίκες που διευκρίνησαν αυτή την τάση, την πολύ σοβαρή του οργανωμένου εγκλήματος ε, τύπου μαφίας που εμπλέκεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δίδεται αυτή η εμπλοκή με την πολιτική. Πολλές χώρες, σε πολλές χώρες είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό τι σημαίνει οργάνωση τύπου μαφίας. Αλλά αυτή η οργάνωση, αυτές οι οργανώσεις δεν αποτελείται από ανθρώπους που ασχολούνται με τις ληστείες μεταφορές κεφαλαίων και ειδικεύονται στην, ε, στο δεθρεμπόριο ναρκωτικών. Οι συνεργάτες της δικαιοσύνης, όταν έγιναν συνεργάτες, ήταν εντός αυτών των, των ε, εγκληματικών οργανώσεων και είπαν μεταξύ άλλων ότι όταν ε, μπαίνουν κανείς σε αυτή την οργάνωση δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Αυτό είναι το σημαντικό πέρασμα. Είναι μια ε, κρυμμένη, μυστική κοινωνία, αν θέλετε, και ομάδα, που ζει από τα έσοδα τα παράνομα και που ουσιαστικά είναι μια κοινωνία ξεχωριστή από την κανονική κοινωνία, που είναι αντίθετη από την ε, κανονική κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει και νομοθετικά να τοποθετηθεί και να αναγνωρίσει νομικά αυτό ε, το έγκλημα της οργάνωσης, της δημιουργίας αυτής της οργάνωσης τύπου μαφίας, ούτως ώστε μετά νομοθετικά να οδηγηθεί σε μια ε, εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Εγώ το λέω αυτό. Και ελπίζω, ε, παρόλο που ήμουν υπερβολικά συνοπτικός, να έδωσα, να κάλυψα όλες τις ερωτήσεις, να έδωσα όλες τις απαντήσεις. Όταν μιλάμε για το ένταλμα σύλληψη. Όταν μιλάμε μετά για την επιχειρησιακή δυνατότητα, εγώ λέω, ναι, λειτουργούμε άριστα. Και με τις νέες χώρες που εντάσσονται και είναι εν ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν υπέροχες, εξαιρετικές σχέσεις. Εμείς οι αστυνομικοί, εμείς οι ερευνητές. Ξέρουμε τη γλώσσα μας μεταξύ μας, είμαστε γρήγοροι, καταφέρουμε να οργανωθούμε. Αλλά μετά όταν βρεθούμε έναντι μηχανισμών θα έλεγα όταν αντιμετωπίζουμε βυζαντινολογίες όπως λέμε στην Ιταλία επιχειρησιακές έχουμε πρόβλημα διότι βρίσκουμε εθνικές νο, ε, νομοθετικές τοποθετήσεις που δεν μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε περαιτέρω τις ερευνητικές μας δραστηριότητε. Ένα απλούστατο παράδειγμα. για, έχουμε πρόβλημα στην Ισπανία για να μπορέσουμε να κατάσχουμε τα έσοδα μια καλαβρέζικη ομάδα. Λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα, τα καταφέραμε, διότι η Ισπανία το κατάφερε. Μέσω μηχανισμών πολύ περίπλοκων βρήκε μια λύση που προβλέπεται από την ομοθεσία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να κατάσχουμε τα αγαθά αυτής της οργάνωσης. Θα πρέπει να βγούμε έξω από αυτή την αμφισημία. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και σαφείς, διότι το οργανωμένο έγκλημα είναι πιο γρήγορο από εμά και πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα και κλείνω με μήνυμα εδώ δεν θα πρέπει να χάσει αυτή την ευκαιρία όπως υπόθηκε με, στην κηδεία του στρατηγού Ντελακέσα. Σε αυτή την περίπτωση μάλλον είπε ο Καρδινάλιος ενώ στη Ρώμη γίνονται συζητήσεις, ε, ε, χάνουμε ανθρώπους. Λοιπόν, λοιπόν, γίνανε πάρα πολλές συζητήσεις, καθυστερήσεις στη Ρώμη και μετά από 8 μήνες έγινε ο φόνος. Λοιπόν, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα συστήματά μας, ούτως ώστε μέσω της εναρμόνισης της νομοθεσίας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε με κοινό μέτωπο αυτού του είδους το, την εγκληματικότητα που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, περίπλοκη εγκληματικότητα και φοβερή διότι ε, είναι σε κρυφή ε, φάση. Στις χώρες όπου δεν υπάρχουν ανθρωποκτονίες, όπου δεν υπάρχουν μηχανισμοί αυτών των βεντετών υπάρχει αυτή η εγκληματικότητα διότι χρησιμοποιεί αυτά που απέκτησε και εξακολουθεί να αποκτά με τη σειρά ετών μέσω ενός από τα εγκλήματα που διαπράττει που είναι το διεθνές ε, λαθρεμπόριο των ναρκωτικών και σταματώ εδώ και ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Διευθυντά Υπάρχουν δύο παρεμβάσεις ε, που ζητήθηκαν. Παρακαλώ να είστε σύντομοι διότι η καθυστέρηση έφτασε 35 λεπτά. Πρώτα ε, ε, κυρία Μπορσελίνο και μετά ο κύριο Δία Δεμέρα για να γίνουν ε, αυτέ οι δύο παρεμβάσει. Ευχαριστώ, λέει κυρία Μπορσελίνο, ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή Αλφόνσο, Αλφόνσο και για το πάθο με το οποίο έκανε την όλη ανάλυση της καταστάσεω και στην Ιταλία και όχι μόνο στην Ιταλία. Από ό,τι κατάλαβα, αυτή η υποτίμηση του φαινομένου ήταν ένα πρόβλημα αρχικά ιταλικό όταν σκεφτόμαστε ότι ε, θεωρώθηκε και ότι η μαφία, η μαφία ήταν πρόβλημα μόνο για την Νότια Ιταλία, αλλά μετά είδαμε ότι ε, εξαπλώθηκε. Και είδαμε και ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Θέλω μια διευκρίνηση από τον κύριο Διευθυντή. Από ό,τι κατάλαβα, η εναρμόνιση του ΣΥΠΗΝ της νομοθεσίας ε, κάποιων στοιχείων είναι η βάση ε, χρειαζόμαστε 416α ευρωπαϊκό να αναγνωρίζετε το έγκλημα παντού. Μας χρειάστηκε πολλής χρόνο αυτός του, το να δημιουργείται μια οργάνωση τύπου μαφίας. Χρειάστηκαν πάρα πολλές φαγές και δολοφονίες για να γίνουν για να το αναγνωρίσουμε αυτό. Θα ήθελα να καταλάβω κάτι. Πιστεύετε κύριε Διευθυντά ότι η παρουσία των μαφιόζικων οργανώσεων στην Ευρώπη είναι μόνο παρακλάδια των νότιων οργανώσεων της Νότιας Ιταλίας μαφία και ντράγκετα ή πιστεύετε ε, ότι ο χώρος στον οποίο εγκαθίστανται αυτές οι, ε, μαφίες είναι, είναι εκεί που υπάρχει δυνατότητα να απτυχθούν, να βλαστήσουν εκ νέου. Δημιουργούνται νέες μαφίες που μοιάζουν, δεν είναι παρακλάδια των αρχικών μαφιών, είναι νέες, μαφ... νέες οργανώσεις που μοιάζουν με τις Ιταλικές μαφίες αλλά έχουν δική τους οργάνωση, δική τους ζωή και δεν εξαρτώνται μόνο από τις αρχικές οργανώσεις, διότι αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Ένα άλλο ερώτημα. Από όταν εφαρμόστηκε το σύστημα της πρόληψης στην Ιταλία, όχι μόνο με την κατάσχεση των αγαθών, αλλά με την κοινωνική χρήση των προϊόντων των κατασχέσεων, κάτι που συζητάμε τώρα στην Ευρώπη υπήρξε μια πραγματική μείωση της εγκληματικής δραστηριότητα ή εξυπηρέτησε μόνο αυτό το μέτρο στην ανάκτηση των αγαθών. Ο κύριος Ντεμέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τη σύνοψη αυτή και κυρίως για το συμπέρασμα. Είναι γεγονός. Οι δημοκρατικές κοινωνίες έχουν ε, υποστεί μια διείσδυση ε, από μαφίες και σε κάποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής τώρα όπου διεισδύουν στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη, στη τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που εξάγεται. Στη χώρα μου, εδώ και πολύ καιρό, ένας δικαστής παίρνει αυτοκίνητα, αεροπλάνα και βαπόρια και τα ε, βάζει ε, στη διάθεση ε, της δικαιοσύνης ένας δικαστής και μόνο για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Ένας δικαστής δίνει εντολή για όλα αυτά τα μέσα για να μπορέσει να καταπολεμά αυτού του είδους τα εγκλήματα. Καλώς, ευχαριστώ. Όταν μιλάω για οργανώσεις τύπου μαφίας. Δεν αναφέρομαι πλέον στην Ιταλία, διότι πιστεύουμε συνολικά ότι η Ντράγκετα, η Καμόρα, η Σάκρα Κορώνα Ουνίτα, η μαφία είναι οργανώσεις που παραδοσιακά αναγνωρίζονται ότι έχουν ρίζες στην Ιταλία. Όχι λιγότερο επικίνδυνες είναι και οι Ρώσικες και οι Κινέζικες οργανώσεις, αλβανικές οργανώσεις. Νιγεριανές οργανώσεις εξάλλου χρησιμοποιούν πρακτικές παράνομες πολύ σοβαρότερες διότι μιλάμε για λαθρεμπόριο ανθρώπων. Πρέπει να πω ότι είναι το φαινόμενο που θα πρέπει να αναλύσουμε εμείς. Συνεπώς είναι ένα πρόβλημα, θα έλεγα ότι σήμερα στην Ευρώπη πέρα από το οικονομικό πρόβλημα, και δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό γιατί δεν είναι αρμοδιότητά μου. Το δεύτερο πρόβλημα όμως, όχι όμως σαν ε, μικρότερη σημασίας, πέρα το οικονομικό πρόβλημα, είναι το εγκληματικό, το πρόβλημα της εγκληματικότητας και αυτή το οργανωμένο έγκλημα. Σήμερα η Ευρώπη, κατά την άποψή μου, ε, ελέγχει καλά το φαινόμενο, το εντοπίζει το φαινόμενο, όταν μιλάμε για την άκτηση των αγαθών, της περιουσίας τους, η ανάκτηση αυτής της περιουσίας είναι θεμελιώδε στοιχείο, διότι παρήγαγε σίγουρα μία ύφεση του φαινομένου της μαφίας, εν γέννη βέβαια, διότι μέσω δύο μηχανισμών το καταφέρουμε αυτό. Μέσω της έκτησης της ποινής, της ποινής με το 41α που προανέφερα και δεύτερο, αυτό που ανέφεραμε. Διότι αυτό δεν είναι τόσο επίκαιρδες το έγκλημα τώρα πια όσο ήταν, διότι όσο γίνεται η ανάκτηση των αγαθών, τους κόβουμε την τροφή, αν θέλετε, από την οποία θρέφεται το οργανωμένο έγκλημα. Όσον αφορά αυτά που έλεγε πριν ο Ισπανός βουλευτής, το επιβεβαιώνω και στην Ιταλία υπάρχει ένας δικαστής ο οποίος κάνει κατάσχεση αγαθών και είπε χρησιμοποιούμε, ε, χρησιμοποιούμε και τα κτίρια. Έχουμε δύο κτίρια ήδη που τα πήραμε το οργανωμένο έγκλημα όπου λειτουργούμε. Τα χρησιμοποιούμε σαν έδρα των επιχειρήσεών μας. Ήδη είμαστε αυτή τη φάση που σίγουρα θα προχωρήσει αυτό και σίγουρα θα οδηγήσει σε αποτελέσματα θετικότατα. Γιατί υπάρχει και ένας κίνδυνος όμως. Πολλές χώρες ευρωπαϊκές, κυρίως της Βόρειας Ευρώπης, δεν έχουν αυτή την οτροπία. Όσον αφορά, δεν αντιλαμβάνονται καλά αυτό του είδους το έγκλημα. Είναι εύκολο να διεισδύσει εκεί η μαφία, αυτές οι οργανώσεις. Γίνεται μια ε, απικιοποίηση, αν θέλετε, των εισαγωγικών. Ε, δημιουργούν απικία αυτοί, αυτές οι οργανώσεις. Και αυτό είναι ο πραγματικός κίνδυνος όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα και διάδοσή του. Ευχαριστώ, Διευθυντά, κυρίω διότι μας δώσατε την εμπειρία σας και κυρίω διότι υπενθυμίσατε ποιοι θα έπρεπε να είναι οι στόχοι και ελπίζω να είναι οι στόχοι αυτής της Επιτροπής σας ευχαριστώ για την ειλικρίνεια και για το πάθος με το οποίο μας μιλήσατε και μας το δώσατε τη γνώση σας και την εμπειρία. Ελπίζω εκ νέου να μπορείτε να ξανάρθετε εδώ για μια μεταγενέστερη συζήτηση όσον αφορά αυτά τα θέματα. Θα δώσω τώρα μέσω το λόγο στο Διευθυντή της Ευρωπόλ, τον κύριο White. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ. Ζητώ συγγνώμη την καθυστέρηση. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να αφαιρέσω το λόγο από κανέναν. Δεν μ' αρέσει να σας στερήσω το λόγο, αλλά σας παρακαλώ να θέσετε ερωτήσεις. Δεν έχουμε χρόνο για να εκφράσουμε σκέψεις. Απλώς ερωτήσεις παρακαλώ, διότι πραγματικά έχουμε ελάχιστο χρόνο. Λοιπόν, κύριε Διευθυντά, από πλευρά Europol και υπό το φως των όσων είπε ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Δαλφόνσο, η αξιολόγηση της Europol για τα διάφορα συστήματα τα εγκληματικά και τη δυνατότητα ε, διάδοσής τους ε, και τι συνέπειε ε, που έχουν όλα αυτά τα συστήματα τα εγκληματικά στην Ευρώπη και τι είναι αναγκαίο κατά την άποψή σα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και να, κάνουμε αυτή τη, να διεξάγουμε αυτή τη μάχη. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε να μιλήσω για τη Europol για το οργανωμένο έγκλημα. Ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη σύσταση τη Επιτροπής σας. Ειλικρινά πιστεύω ότι χρειαζόταν εδώ και πολύ καιρό και θεωρούσα ε, εδώ και καιρό ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πιο εστιασμένη προσέγγιση και πιο μεγαλύτερη συγκέντρωση στο οργανωμένο έγκλημα, διότι επηρεάζει τόσους πολλούς πολίτες στην Ένωση. Θα ήθελα να καλωσορίσω αυτό το βήμα και ε, το υποστηρίζει πολύ η Europol και θα πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε διατεθειμένοι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε το επόμενο έτος στην Επιτροπή σας. Ποιος είναι ο στόχος? Να επικεντρωθείτε σε αυτό που έχουν σημασία στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι μια πολιτική και ένα περιβάλλον πολύ περίπλοκο και σύνθετο και αφορά περισσότερο κλάδ, περισσότερους κλάδους της κοινωνίας από όσο νομίζει ο κόσμος γενικά και έχει και πολύ ισχυρό πλαίσιο πολιτικής που συνδέεται με αυτό στο νέο κύκλο καταπολέμησης του οργανωμένου κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί το Κοινοβούλιο να δυναματίσει ιδιαίτερο ρόλο και να επικεντρωθεί σε τομείς κλειδιά αυτού του προβλήματος. Αλλά είναι μεγάλη πρόκληση για σας κυρία Πρόεδρε πιστεύω για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε πραγματικά να εστιαστείτε στα σημαντικά και τι μπορεί να φέρει ως προστιθέμενη αξία το Κοινοβούλιο σε αυτή τη σημαντική συζήτηση. Η Europol έχει να παίξει εδώ ιδιαίτερο ρόλο και βεβαίως βοηθούμε τις αρχές των κρατών μελών να καταπολεμούν το έγκλημα πάνω από μία εικοσαετία από τη στιγμή που συσταθήκαμε. Πάντως εδώ η πρωτογενής δράση και η βασική παραμένει φυσικά άμεσα στα κράτη-μέλη. Το αναγνωρίζουμε αυτό το γεγονός. Η Europol εδώ δεν έχει έρθει για να αναλάβει αυτή την ε, αρμοδιότητα και την ευθύνη, αλλά για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να δώσει την υποστήριξη που χρειάζονται για να καταπολεμούν το έγκλημα αποτελεσματικά. Κατά αυτή την 20 ετία λοιπόν που ε, εργαζόμαστε, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη. Ε, δεν ήταν εύκολο, δεν πετύχαμε τα πάντα έχουμε όλο και περισσότερες επιτυχίες επιχειρησιακές και περισσότερες ευθύνες ε, ε, μας δίνουν οι ε, αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής και μπορούμε από κοινού να καταπολεμούμε το έγκλημα. Έχουμε πολύτιμη εμπειρία σε κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος αλλά και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. 800 περίπου είναι το προσωπικό μας στη Χάγη, στα νέα μας κτίρια, στην έδρα μας, από κάθε υπηρεσία στην Ευρώπη που έχει να κάνει με οποιαδήποτε μορφή κλιματικής δραστηριότητας. Ε, έχουμε 150 συνδέσμους αξιωματικούς, ε, επιχειρησιακούς, άνδρες και γυναίκες από τα κράτη-μέλη και από αλλού στην Ευρώπη που συνεργάζονται στα κτίρια μας ε, στεγάζονται μαζί και χρησιμοποιούν ε, τη βάση δεδομένων μας κάθε μέρα. Είναι πραγματικά ένας λιμένας επιχειρησιακός δράσης, ε, μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη ως περιβάλλον επιχειρησιακής λειτουργίας και κέντρου και κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε. Αυτή η κοινότητα λοιπόν επιχειρησιακών ε, ε, υπαλλήλων και αναλυτών ε, κάνει 14.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αυτό αφορά τις πιο επικίνδυνες εγκληματικές οργανώσεις και τρομοκρατικές οργανώσεις. Ζητήθηκε, μου ζητήθηκε να σας εξηγήσω ε, το ιδιαίτερο πρόβλημα της Ιταλικής μαφίας ακούσαμε προηγουμένως και πώς ε, παραμένει απειλή για την ασφάλεια όχι μόνο της Ιταλίας αλλά και ε, της υπόλοιπης Ευρώπης. Συμφωνώ. Φαίνεται αυτό από την επιχειρησιακή δουλειά που κάνουμε και από τις εκτιμήσεις μας. Αλλά είπαν και άλλοι. Εγώ άκουσα την ερώτηση της κυρίας Μπορσαλίνο. Είναι διάφορες οι παράμετροι και οι μεταβλητές του προβλήματος της μαφίας, για να το χαρακτηρίσω έτσι, σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Αλλού βλέπουμε αυτές τις οργανώσεις οικογενειακού τύπου, εγκληματικέ οργανώσεις, ενώ σε άλλα μέρη έχουν διαφορετική δομή και οργάνωση. Είναι πιο δυναμική και πιο ρέουσα, δεν ε, απορρέει από μέλη της ίδιας οικογένειας ή την ίδια εθνότητα, αλλά ε, διαπερνά διάφορες εθνότητες και ε, κρατικά σύνορα. Το συνδικάτο του εγκλήματος, ε, ας πούμε, από κάποιο μέρος της Ευρώπης που απλώνει τα πλοκάμια του σε πολλούς κλάδους και μέχρι την νόμιμη οικονομία. Και στην Ευρώπη αυτό το βλέπουμε. Είναι πολύ υψηλή ευελιξία τους, η δυναμική τους, ε, εκμεταλλεύονται τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή, εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, ε, όπως έχουμε σήμερα, για να εκμεταλλεύονται πολίτες, εταιρείε και κυβερνήσεις ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι μια εικόνα οργανωμένου εγκλήματος με διαφοροποιημένη φύση, ε, η παραδοσιακή μαφία και το πρόβλημά της είναι ένα σκέλος. Σημαντικό μεν, αλλά ένα μόνο. Ε, και μία από τις διαστάσεις και τις εκδηλώσεις και εκφάσεις του προβλήματος. Πού φαίνεται αυτό. Οχτώ είναι οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες στην Ευρώπη. Οχτώ για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το κυβερνοέγκλημα είναι ένα, αλλά και άλλες σημαντικές διαστάσεις σε ποιο βαθμό τα Βαλκάνια παραμένουν πολύ σημαντικοί ε, ε για αυτές τις δραστηριότητες. Η Δυτική Αφρική, ας πούμε, για το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και τη διακίνηση ανθρώπων, δουλεμπόριο. Εδώ και χρόνια στη Europol εκτιμούμε αυτά και σε αιτήσια βάση ε, εκδίδουμε από το 2006 τα συμπεράσματα. Επιτρέψτε μου να καλύψω μερικές από τις βασικές τάξεις. Ε, αυτές οι ευέλικτες ομάδες λειτουργούν σε διάφορες εθνικές δικαιοδοσίες και πάλι βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ διαφόρων ε, εθνικοτήτων. Οι Αλβανόφωνοι, ας πούμε, οι Λιθουανοί είναι οι πιο οργανωμένοι, ε, αλλά και εκείνη της Ιταλίας τώρα έχουν πολύ διαφορετικές δραστηριότητες και χαρτοφυλάκια. Ε, επίσης, ε, ε, υποπτευόμαστε ότι συνεργάζονται και περισσότερο με τη τρομοκρατία σε ορισμένους τομείς και χώρους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων και τρομοκρατίας. Στο μεταξύ, έχουμε και νέο είδος ε, παραποίησης ε, πιστοτικών ε, καρτών, συγγνώμη, χρεωστικών καρτών και παραποίηση και πλαστογράφηση εμπορευμάτων και στο διαδίκτυο, γιατί ακόμα ο νομοθέτης δεν έχει προλάβει να τα ρυθμίσει αυτά και είναι χαμηλότερη και η κίνδυνη και χαμηλότερα και τα πρόστιμα που συνδέονται με αυτές τις δραστηριότητε. Παρ' όλα αυτά, ε, είναι πολύ μεγάλη ζημιά και στην οικονομία και στους πολίτες μας. Παράδειγμα, πρόσφατα στην Ισπανία χωροφυλακή ε, ε, το Μάρτιο σε συνδυασμό με τη Europol και τη συμμετοχή και άλλων κρατών μετών βρήκε 30.000 δόσεις πλαστών φαρμάκων και τις κατήσχε. Αυτό ε, αφορούσε πολύ μεγάλες ποσότητες πλαστών φαρμάκων. Είναι μια νέα διάσταση που αντιμετωπίζουμε και συγκεκριμένη και ιδιαίτερη ζημία στους πολίτες. Επίσης βλέπουμε μια τάση ε, σε δραστηριότητες όπως είναι η παραχάραξη νομισμάτων πιο συχνά ε, για να χρηματοδοτήσουν άλλου είδους παράνομες δραστηριότητες όπως είναι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Επίσης χρησιμοποιούν και κοντέινερ αλλά και επιβατηγά πλοία και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελέγξει κανείς ως προς την ασφάλεια των συνόρων αυτή την κυκλοφορία και το εμπόριο και τον όγκο απλούστατα ε, κοντέινερ που κυκλοφορούν κάθε μέρα στη θάλασσα. Είναι τεράστιο το δίκτυο των ναυτικών και των θαλασσίων μεταφορών. Δεν μπορεί κανείς να ελέγχει ε, όλα αυτά τα πλοία που μπαίνουν σε τόσα πολλά λιμάνια στην Ευρώπη σε καθημερινή βάση αυτό μπορεί να γίνει μόνο με πολύ καλή πληροφόρηση και στοχευμένη. Ακόμα και οι οδοί έχουν αλλάξει και έχουν γίνει πιο δυναμικές σε σχέση με το παρελθόν. Όπως σας είπα, η Δυτική Αφρική χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά για τη διαμετακόμιση και διάφορα τα σημεία εισόδου και διαφορετικά ανάλογα με το προϊόν, κοκαίνη, ηρωίνη κτλ. Το έχουμε δει και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ροές λάθρομεταναστών και δουλεμπόρων. Έχουμε λοιπόν ε, μια νέα κατάσταση και θα πρέπει η Ένωση να δραστηριοποιηθεί, να έχουμε πιο συντονισμένη δράση, ακόμα περισσότερο και όχι λιγότερο. Όπου υπάρχει βασική ευθύνη για εφαρμογή ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο και βέβαια αυτό παραμένει στα κράτη των κρατών μελών, δεν χωράει καμιά αμφιβολία, αλλά μόνα τους δεν μπορούν να δράσουν. Θα πρέπει να είναι ένα τμήμα μιας συντονισμένης και ενιαίας απάντησης κατά πολέμηση του εγκλήματος και της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μία από τις πρώτες αποστολές θεσμών όπως είναι η Europol. Να έχουμε πιο αποτελεσματική ε, απάντηση σε όλη την Ευρώπη και σε όλες τις προκλήσεις του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Αναφέρθηκα ε, την ιδιαίτερη επίπτωση στην οικονομία. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα, έτσι όπως είναι κρυμμένο, συχνά ε, έχει διστήσει στην οικονομία και ε, επηρέαζε και την Ένωση στη δυνατότητά της να αντιμετωπίσει την παγκόσμια κρίση. Ε, είναι πιο βάλωτη ε, η κατάσταση στη διαφθορά. Οι μεγάλες διαφορές στο ΦΠΑ που είναι πάνω από 100 δις ευρώ το χρόνο. Αυτό το εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο οργανωμένο έγκλημα, στο πώς προσαρμόζεται ε, στην επιγραμμική απάτη. 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά βγαίνουν από την νόμιμη οικονομία ακριβώς τη στιγμή που οι εθνικές κυβερνήσεις το χρειάζονται για να μειωθεί το χρέος τους και για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την ανάκαμψη της οικονομίας. Να, μην γελιέστε, υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ της δυνατότητας των κυβερνήσεων να εξασφαλίσουν την οικονομική ανάκαμψη και ε, τις δράσεις οργανωμένου εγκλήματος σήμερα στην Ευρώπη. Λατρεμπόρι τσιγάρων κοστίζει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και πάλι αυτά είναι χρήματα ε, θεμητά και νόμιμα φορολογικά έσοδα που εκφεύγουν του κράτους. Ε, αυξάνεται η ανεργία και ε, τα άτομα είναι πιο ευάλωτα στην πρόσληψη του στρατολόγηση από εγκληματικές ομάδες. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε, να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα σε όλες του τις εκφάνσεις στην Ευρώπη. Θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους ίδιους τους εγκληματίες ότι εμείς είμαστε ισχυροί, ισχυρότεροι απέναντί τους και στις νέες απειλές. Θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες ότι από κοινού συνεργαζόμαστε όσο μπορούμε, όσο σκληρά μπορούμε για να τους προστατεύσουμε τις νέες απειλές και στη Ένωση ε, και σε κλειστούς χώρους αλλά και στους δρόμους, στους δημόσιους χώρους. Το κυβερνοέγκλημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αυτό θα το συζητήσουμε αργότερα και εσείς στην Επιτροπή σας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εκτιμάται ότι είναι εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα ευρώ που χάνουν κάθε χρόνο οι επιχειρήσεις. Εργαζόμαστε πολύ σκληρά στη Europol και στον τομέα αυτό και χαιρόμαστε πολύ ε, από τη δραστηριότητα που έχουν αναλάβει και η Υπουργή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συσταθεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκκλήματος το 2013 στην Europol. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και πιστεύουμε ότι θα είναι πραγματικά κομβικό σημείο της απάντησης της Ένωσης ε, στο κυβερνό έγκλημα. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό για να ε, κλείσουμε αυτές τις νέες πόρτες που ανοίγουν οι εγκληματίες για να κάνουν κακό στην κοινωνία. Και καμιά φορά ε, παίρνει και ουσιαστική μορφή αυτό. Εκατοντάδες θύματα ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών κάθε χρόνο ε, εντοπίζονται και... Το οργανωμένο έγκλημα λοιπόν βλέπετε ότι έχει μια παλέτα δραστηριοτήτων, δεν είναι κοινή. Αυτό που βλέπουμε στην Ιταλία δεν είναι το ίδιο με αυτό που σημαίνει στη Λιθουανία, για παράδειγμα, ή αλλού στη βόρειο-ανατολική Ευρώπη, ή αυτό που βλέπουμε να συμβαίνουν, ε, ξέρω εγώ, στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι τέσσερις ή πέντε οι τομείς, τα επίκεντρα ε, οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη, σε αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα, και είναι η βασική κόμβη ε, λειτουργία του οργανωμένου εγκλήματος και ενδεικτική για το πώς διανέμονται τα λαθρέα εμπορεύματα, ε, πώς ε, συναντώνται για να συντονίσουν τις δραστηριότητες τους οι ομάδες αυτές, για ποιο τρόπο χρηματοδοτούνται και επίσης πώς διοχετεύουν τα χρήματα αυτά και πώς τα ξεπλένουν και μπαίνουν στην πραγματική οικονομία. Λοιπόν, υπάρχουν βασικοί κόμβοι στην Ευρώπη και είναι σημαντικό από κοινού να τους χτυπήσουμε αυτούς τους κόμβους πάρα πολύ ε, αμήλικτα. Βεβαίως γίνεται εξαιρετική δουλειά στην Ιταλία για την καταπολέμηση της μαφίας εκεί, αλλά ε, δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τις άλλες περιοχές που σας ανέφερα. Τι θα πρέπει να γίνει τώρα. Προσωπικά σας είπα και πριν, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή για να είμαστε και πιο ισχυροί εν τη ενώση για να καταπολεμούμε το οργανωμένο έγκλημα. Στη Europol εμείς είμαστε οι μεσολαβητές, οι διευκολυντές ας πούμε, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας να δράσουμε. Ε, είμαστε υποχρεωμένοι να επαφιέμεθα στα κράτη-μέλη. Και στο νέο κανονισμό αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη-μέλη. Αν δεν έχουμε πληροφορίες, δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε τις δραστηριότητες, να τους ξεσκεπάσουμε. Θα πρέπει να βρούμε ένα ευφυή τρόπο να δίνουμε κίνητρα στις διοκτικές αρχές των κρατών μελών, πολλές φορές να σκεφτούνται πιο ευρωπαϊκά και λιγότερο εθνικά γιατί σε κάθε μεγάλη δίωξη και έρευνα που γίνεται σε εθνικό επίπεδο σίγουρα υπάρχει διεθνής διάσταση που υπερβαίνει τη δικαιοδοσία του κράτους μέλους. Και μέχρι στιγμής η νοοτροπία, η κουλτούρα των διοκτικών αρχών είναι εθνική και αυτό δεν έχει αρκετά εξυγχρονιστεί για να αντιμετωπίσει την ευρωπαϊκή και τη διεθνή διάσταση με τον τρόπο που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Εμείς μετά από 20 χρόνια στη Europol εξυγχρονίζουμε τις εγκαταστάσεις, τις υπηρεσίες, εσωτερικά να διοργανόμαστε. Ε, ε θα έχουμε το κέντρο για την καταπολέμηση του κυβερνού εγκλήματος. Ένας από τους ε, τρεις βασικούς τομείς. Οι άλλοι δύο είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Οργανωμένο έγκλημα εστιάζουμε και στην Ιταλική μαφία και μαζί με τους Ιταλούς και άλλους κάνουμε εκτιμήσεις για τον κίνδυνο, για πώς έχει η ευρωπαϊκή εικόνα αυτού του προβλήματος. Αλλά επίσης δραστηριοποιούμαστε και σε άλλους τομείς που μας ανησυχούν. Από την Ανατολική και Βόρεια Ευρώπη υπάρχουν ομάδες πάρα πολύ ευκίνητες που δρούν σε τουλάχιστον 20 χώρες. Και αυτό εμφανίζεται επίσης και στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι ε, όλα αυτά ε, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Δεν είναι μόνο η φωνή του λαού και η δημοκρατική νομιμότητα, αλλά και κάτι ακόμα. Υπάρχει ένα αίτημα να βοηθήσει το Κοινοβούλιο σε, αυτό που είπε ο Διευθυντής Ταλφόνσο, να καταλάβει ο κόσμος, το κοινό, ότι είναι σημαντικό να μην υποτιμάτε το έργο του οργανωμένου εγκλήματος. Ότι το χέρι του οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται ότι έχει μπει σε πολλούς τομείς της κοινωνίας, τις επιχειρήσεις, πώς λειτουργούν, πώς τρευλώνεται ο ε, ανοιχτός και υγιής ανταγωνισμός στην αγορά, πώς διανέμουν ναρκωτικά σε κάθε μεγάλο πολίτη της Ευρώπης και όχι μόνο και σε κάθε γωνιά του κάθε δρόμου. Ε, νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει διανοηθεί, δεν έχει αντιληφθεί ε, και κατανοήσει καλά τι συμβαίνει. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ε, στον κόσμο, στην κοινωνία. Επίσης το Κοινοβούλιο ως Δημοσιονομική Αρχή έχει και την ευκαιρία να βεβαιωθεί ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητοι πόροι γιατί σε τελική ανάλυση πρόκειται για παράνομη οικονομία που ε, οδηγεί σε απώλειες δισεκατομμυρίων ευρώ από τους προπολογισμούς μας. Και από τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε ε, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε καλύτερα τους ε, θεσμούς και τις οργανώσεις που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Και τέλος, η Europol θα υποστηρίξει οπωσδήποτε τις ε, εργασίες της Επιτροπής σας. Ε, προσβλέπω ε, στη δική σας συνεισφορά και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Ελευθεριών στα πλαίσια της αναθεώρησης του κανονισμού μας. Είμαστε πραγματικά ευγνώμονες για την υποστήριξη που θα μας στείλετε για να υπάρχουν μεγαλύτερα κίνητρα για τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται καλύτερα με την Europol, να υπάρχει ένα ε, πιο σύγχρονο σύστημα ανάλυσης και αποθήκευσης των στοιχείων. Σε ό,τι αφορά το πώς εμείς μπορούμε να σας υποστηρίξουμε, σας είπα και στην κυρία Αλφάνο ότι μπορεί 100% να υπολογίζει στη δική μας υποστήριξη, θα φέρω στην Επιτροπή σας μάλλον θα σας διαθέσω ένα μόνιμο εμπειρογνώμονα για να σας υποστηρίζει σε ειδικού τομείς όπου χρειαστείτε. Οι απειλές και οι εκτιμήσεις τους, ε, σας είπα, είναι κάτι που μας απασχολεί και θα σας τα διαβιβάζουμε και σε εσά. Έχετε την πλήρη υποστήριξή μας, τον πλήρη σεβασμό μου ε, για τη σημασία που δίνει πλέον το Κοινοβούλιο σε αυτό το σημαντικό τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά διότι είπατε εκ νέου ότι είσαστε διαθέσιμος για τις συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι χρειάζεται να γνωρίζουμε και να κατατήσουμε ένα σχέδιο δράσης και χρειάζεται η άποψη των ειδικών, η δική σας και κυρίως η υποστήριξή σας. Και τώρα δίνω το λόγο στις ομάδες για ένα δίλεπτο και όχι παραπάνω. Αλλιώς θα είμαι υποχρεωμένος να σας φέρω στο λόγο. Η κυρία Ματιό έχει το λόγο. Ευχαριστούμε τον κύριο Γουένου Ράιτ για αυτή την πλήρη παρουσίαση που πραγματικά μας προβληματίζει βλέποντας την εξέλιξη αυτού του οργανωμένου εγκλήματος. Μια κοινωνία μέσα στην κοινωνία μας. Μας φοβίζει αυτή η εξέλιξη. Δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τα μέσα, τα επιχειρησιακά και τα νομικά για να πολεμήσει κανείς αυτή την εξέλιξη, αυτή τη μαφία. Και ελπίζω ότι αυτή, η σύσταση αυτής της Επιτροπής θα μπορέσει να σας βοηθήσει στο τέλος των εργασιών να πολεμήσετε το οργανωμένο έγκλημα. Και λυμάμαι που ο προϋπολογισμός ε, από χρόνο σε χρόνο δεν βρίσκεται στο επίπεδο που χρειάζεται για να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα. Ελπίζω επίσης ε, το κέντρο για το έγκλημα αυτό κυβερνοχώρο ε, ελπίζω λέω γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν θα υπάρχουν τα διαθέσιμα, οι διαθέσιμα μέσα για να μπορέσει κανείς να λειτουργήσει σε αυτή την ενότητα. Τώρα, για τη διάδραση ανάμεσα, στις, ανάμεσα στη τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα. Είπατε ότι κάποιο θέμα χρηματοδότησης υπάρχει σε αυτούς εδώ τους δύο χώρους. Θα ήθελα να ξέρω λίγο περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κυρία Μάτιε κ. Μίνσκι έχει το λόγο. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Για το θέμα αυτό θα ήθελα να πω ότι ευχαριστώ τον κύριο Ράιτ για τις πληροφορίες που μας έδωσε. Κύριε Ράιτ, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ότι σήμερα το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει την ίδια επιρροή όπως πριν από 20 χρόνια, τουλάχιστον στη Λετωνία. Πριν από 20 χρόνια είχαμε συμμορίες. Δεν τις έχουμε πια. Δεν έχουμε τόσες πολλές μάλλον. Εγώ εργάστηκα στην ε, αστυνομία που καταπολέμησε αυτούς του είδους τις ομάδες και γνωρίζω. Σήμερα η διαφθορά είναι το σοβαρότερο πρόβλημα και οι συνέπειες της διαφθοράς είναι πραγματικά καταστροφικές. Θα πρέπει να εστιαστούμε επί της καταπολεμήσεως της ε, διαφθοράς Δυστυχώς η Λετωνία αντιμετωπίζει βαθιά κρίση αυτή την εποχή και το οργανωμένο, το οργανωμένο έγκλημα με τη διαφθορά είναι πολύ ισχυρό και μπορεί να υπονομεύσει το ίδιο το κράτος. Πέρσι το κοινοβούλιο της Λετωνίας διαλύθηκε λόγω σκανδάλου διαφθοράς πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά πολεμήσεως της διαφθοράς, πρέπει να αναλυφθούν σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Το οργανωμένο έγκλημα γίνεται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και είναι σχεδόν αδύνατο μια χώρα μόνη της να το καταπολεμήσει. Αν η συνεργασία μεταξύ των χωρών είναι ανεπαρκής, τι μηχανισμούς έχει στη διάθεσή σας για να πετύχετε το στόχο σας. Αυτή είναι η ερώτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για την Άλτε, δύο λεπτά, ο κύριος Νιούτον Ντόν. Ε, κύριε Διευθυντά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πολλά πράγματα που δεν είχατε χρόνο να μας αναφέρετε και προσβλέπουμε σε μελλοντική συνεργασία. Στο τέλος είπατε και συμφωνώ με αυτό εκβαθέων ότι είναι θέμα ενημερώσεως του κοινού. Αν μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για την κλίμακα του προβλήματος θα εξοργιστούν και θα τεθεί η πίεση επί των εθνικών ηγετών να κάνουν κάτι. Άρα θα πρέπει να κινητοποιήσουμε το κοινό και θα ακολουθήσουν οι ηγέτες. Αυτή είναι η απλή πολιτική διαδικασία. Δεν λειτουργεί, ε, δεν κινούνται οι ηγέτες αν δεν δεχτούν πίεση και αυτό θα πρέπει να κινητοποιήσουμε. Έχω πολλές ερωτήσεις, αλλά θέλω να πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που είπατε, τα 4-5 επίκεντρα του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη. Ίσως είδα πολλές ταινίες του James Bond αλλά δεν μπορώ να φανταστώ αυτές τις τεράστιες επιχειρήσεις να λειτουργούν πάρα πολύ ευέλικτα με την πρόσφατο εξοπλισμό και τους πιο πρόσφατους υπολογιστές εκτός αν κάπου υπάρχει κάποιο κτίριο το οποίο υπάρχουν και εργάζονται. Αυτός ο επικεφαλής, ο κ. Μπίκ δεν έχει κάπου ένα γραφείο. Τέσσερις-πέντε ουρανοξύστες στην Ευρώπη, σε κάποια μέρη της Ευρώπης όπου η, διεθ... διεθνής εγκληματικότητα ΑΕ εργάζεται δεν πρέπει να είναι μόνο σε σπίτια. Μια εικόνα δεν μπορείτε να μα ζωγραφίσετε πώ περίπου λειτουργεί το όλο σύστημα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κύρκοπ έχει το λόγο τώρα. Του συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ, ε, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον κύριο Γουέιν Ράιτ. Τον έχουμε δει επανειλημμένα στο παρελθόν. Πάρα πολύ μα βοήθησε και στην νομική επιτροπή ιδιαίτερα ε, για το έργο της Europol. Έχω δύο σημεία ερωτήσεις σύντομα, Πρόεδρε. Πρώτον, συζητήσαμε για τις εξουσίες ε, Europol στο παρελθόν επανειλημμένα. Εγώ έχω εκφράσει τις απόψεις μου. Υπάρχουν ένα-δύο τομείς που θεωρώ ότι θα ενδιέφεραν τη Europol να ασχοληθεί ακριβώς λόγω των διοργανικών σχέσεων. Δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Θα ήθελα να ρωτήσω τι λέει ο κύριος Γουάινραϊτ, ε, θα τον βοηθούσε και στο δικό του έργο και στη δική μας επιτροπή στην καταπολέμηση της μεγάλης εγκληματικότητας. Εάν είχατε περισσότερες ε, εξουσίες και αν ποιες ε, θα ήταν αυτές. Και δεύτερο, Θέλω να πω το εξή για να γραφτεί και στα πρακτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η Επιτροπή και συστήθηκε για να αντιμετωπιστεί μια πολύ σοβαρή κατάσταση στην Ευρώπη με το οργανωμένο έγκλημα και γι' αυτό εκπλήσωμαι, δεν φαντάζομαι θα μπορέσει να το σχολιάσει αυτό, για τις δράσεις του δικού μου κοινοβουλίου που σταμάτησε ε, τις ε, διαπραγματεύσεις για το κυβέρνο έγκλημα, για την Ευρωπαϊκή Εντολή ε, Σύλληψης και για την έκθεσή μου για το PNR το ίδιο αυτό το τόσο κρίσιμο ε, καιρό για τις τύχες μας που είναι τόσο σημαντική η ασφάλεια για όλους μας. Το PNR είναι η λύση με τα δεδομένα των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Ε, ε, φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να απαντήσει, δεν περιμένω να απαντήσει, αλλά να γραφτεί στα πρακτικά, Πρόεδρε, ότι αυτές είναι οι απόψεις μου σήμερα το πρωί σαφέστατες. Σας ευχαριστώ. Δύο λεπτά, κύριο Σόντεργκατ, για την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας. Έχω μία-δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα έχω να ρωτήσω το εξή. Ο κ. Διευθυντής αναφέρθηκε στο θέμα του εμπορίου ανθρώπων. Θα ήθελα να γνωρίζω λίγα κάποια περισσότερα πράγματα για αυτή την πτυχή ε, όσον αφορά το εμπόριο σαρκός που σχετίζεται και με την παράνομη εργασία. Ε, η Δανία, στη Δανία βλέπετε ότι όλες οι μεγάλες αξιοσέβαστες κατασκευαστικές εταιρείες και οι σεβαστές εταιρείες καθαρισμού, αν εξετάσετε υπεργολαβίες και λοιπά και το ψάξετε κάπως, βλέπετε ότι η αγορά εργασίας που κινείται εκεί είναι παράνομη, δεν καταβάλλονται φόροι ε, και μεγάλα ποσά αφορούν τη φοροδιαφυγή και αυτοί που εργάζονται, ε, εργάζονται σαν δούλοι. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα όσον αφορά αυτή την πτυχή και τι ρόλο παίζουν αυτές οι επιχειρήσεις σε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. Δεύτερον ερώτημα. Είπατε ότι σε όλες τις μεγάλες έρευνες σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα υπάρχει και μια διεθνής διάσταση. Συμφωνώ με αυτό. Θα ήθελα να ξέρω αυτό είναι μόνο ευρωπαϊκό φαινόμενο, ευρωπαϊκή διάσταση ή διάσταση που ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης. Θα ήθελα να μας πείτε και κάτι για τη σχέση μεταξύ Europol και Interpol. Διότι αν η διεθνή διάσταση ξεπερνά την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν χρειαζόμαστε μόνο στενότερη συνεργασία σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επίπεδο Interpol. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τον κύριο Wainwright, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Wainwright, να σα ρωτήσω κάτι. Πολύ συχνά μιλήσαμε για του στόχου τη Επιτροπή και πάνω απ' όλα για το πώ μπορεί αυτή η Επιτροπή να συμβάλλει σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Είναι και μια ιστορική ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην παρέμβασή σας σωστά υπογραμμίσατε επανειλημμένα συνεργασία και σύμπραξη. Αυτές είναι βασικές εκφράσεις, λέξεις κλειδιά. δεν υπάρχει ένα μέρος που να, ε, να μην πάσχει από, την, ε, από το οργανωμένο έγκλημα. Στα 27 κράτη-μέλη δεν υπάρχει μια περιοχή, ένας χώρος που θεωρείται ασφαλής. Διότι είναι τόσο μεγάλα τα συμφέροντα βέβαια. Έχουμε τη διαφθορά. Ε, το ξέπλυμα χρήματος. Λυσμονούμε πολύ συχνά τότος το συμφέρον που έχουν αυτά τα εγκληματικά συστήματα. Αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εδώ και κάποια χρόνια ε, μία από τις εγκληματικές οργανώσεις, τις πιο προχωρημένες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον κόσμο, μπόρεσε να ανακυκλώσει, αν θέλετε, να ξεπλύνει σε μία μέρα στο Βέλγιο, εδώ, 28 εκατομμύρια ευρώ. Σε μία μέρα. Και το ξέρουμε αυτό διότι εντοπίστηκε. Πόσες όμως άλλες τέτοιες πράξεις μας ξέφυγαν και πόσα άλλα χρήματα ε, ξεπλήθηκαν σε μια μέρα. Πιστεύω δεν λάβαμε ίσω υπόψη το πώς εξελίχθηκαν αυτές οι οργανώσεις εκμεταλλευόμενες την άγνοια και την αδιαφορία ε, κάποιων κρατών μελών όσον αφορά τα προβλήματα. Ε, νομίζω ότι πρέπει πραγματικά να έχουμε το σωστά μέσα στη διάθεσή μας. Η Europol θα πρέπει να ενισχυθεί. Θα πρέπει να πιστέψουν τα κράτη μέσα στη Europol διαφορετικά ε, πώς να εφαρμόσουμε τη συνεργασία. Θα ήταν μάταιοι θα παίζα είναι σαν ένα παιχνίδι που το παίξαμε μόνο μέχρι το ημίχρονο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις πολύ καλές ερωτήσεις και παρατηρήσεις που κάνατε για την τρομοκρατία και το οργανωμένο κλίμα. Νομίζω ότι τα στοιχεία δεν είναι ακριβώς πιστικά. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και προσελκύει πολλούς σχολιαστές να το ε, σχολιάζουν. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο 100% ότι υπάρχει πάρα πολύ ισχυρή διασύνδεση, αλλά ορισμένα στοιχεία μα ανησυχούν από αυτά που παρατηρούμε. Είδαμε παραδείγματα στη Δυτική Αφρική. Ε, Η εισαγωγή ναρκωτικών χρησιμοποιείται για την άμεση χρηματοδότηση ε, τρομοκράτες που συνδέονται με την Αλκάιντα και δρούν σε διάφορα μέρη της Αφρικής και ε, από διάφορα μέρη της Αφρικής και διεθνώς. Τα στοιχεία ακόμα όμως δεν είναι ε, κάτι που μπορούν να μας οδηγήσουν σε βάσιμες υπόνοιες, αλλά μας κάνουν να ανησυχούν. Για το σχόλιο τώρα σχετικά με την πρόοδο που έχει γίνει στη Λετωνία. Τον περασμένο μήνα πήγα στη Λετωνία και είδα τον εθνικό ε, επιθεωρητή, τον κύριο Κούζης, κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχει μειωθεί πολύ ε, η χρηματοδότηση της αστυνομίας λόγω οικονομικών προβλημάτων της χώρας. σε ε, πολλά μέρη της Ευρώπης δεν βλέπουμε ένοπλες συμμορίες στους δρόμους, αλλά αυτό έχει αντικατασταθεί από πιο εικονικά όπλα. Ας πούμε, υποκλοπή και παραποίηση ταυτότητας ε, ε, για να τρομοκρατούν και να εκφοβίζουν τον κόσμο πολύ περισσότερο από ό,τι πριν από 20 ή 30 χρόνια. Πλαστοπροσωπεία δηλαδή και στους δρόμους και στη Λετωνία και αλλού μπορεί να έχει μειωθεί η απειλή, αλλά βλέπουμε άλλους τρόπους ε, πιο ύπουλους και δόλιους που εκτείνονται σε μεγαλύτερες επικράτειες και με τρόπο πιο ομοιόμορφο από ό,τι βλέπουμε μέχρι σήμερα. Σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, το ανέφερε ο κύριος Νιούτον Ντάν, το είπα και εγώ. Πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται περισσότερο την απειλή από την τρομοκρατία παρά το οργανωμένο έγκλημα. Είναι γεγονός αυτό, αλλά είναι αναντίστοιχο. Το οργανωμένο έγκλημα βλάπτει πολύ περισσότερο τους πολίτες από οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατίας. Βέβαια δεν υπάρχει μια ευθεία αναλογία, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουν και εκείνοι που χαράσουν πολιτική. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ε, ε, πολλά κτίρια του κυρίου Big ή του κυρίου Μεγάλου. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια και τόσοι μεγάλοι. Στην Ιταλία ε, υπάρχουν άλλοι εμπειρογνώμονες και ξέρουν καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχει ακόμα αυτή η φιγούρα ε, του νονού, αλλά δεν υπάρχει πια τόσο μεγάλη ιεραρχική δομή. Ε, είναι πιο μικρές οι ομάδες και έχουν τις έδρες τους εικονική μορφή και δρούν με έναν τρόπο πολύ πιο αόρατο, δυσδύοντας την οικονομία. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Συμφωνώ με τον κύριο Κίρκοπ. Περισσότερες εξουσίες για τη Europol μπορεί να μας βοηθάει αυτό το καιρό. Η συνθήκη της ίδια ξεκαθαρίζει ποια είναι τα φυσικά όρια ε, των αρμοδιοτήτων της Europol και δεν θα πρέπει να εξελιχθεί και να γίνει ένα όργανο ή μια υπηρεσία με εκτελεστικές εξουσίες. Θα πρέπει να είμαστε πιο ευφυείς και να επικεντρωθούμε στην πραγματική ε, αξία και μοναδική αξία της Europol. Το είπε η κυρία Αλφάνο προηγουμένως. Ε, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη συνεργασία και τη σύμπραξη και σε επιχειρησιακό επίπεδο να βελτιώσουμε την κοινή μας απάντηση στο έγκλημα στην Ευρώπη. Να χρησιμοποιείται η Europol ε, ως το κέντρο ενημέρωσης που είναι για την καταπολέμηση. Να ενισχύσουμε κοινέ ε, προδιαγραφές και πρότυπα ε, στα κράτη-μέλη. Να ενισχύσουμε τα βασικά εργαλεία για το κυβερνό έγκλημα, για το ξέπλυμα χρήματος. Όλα αυτά είναι κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία στη Europol που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο για την επιχειρησιακή δράση στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή. Αυτό το όραμα έχω εγώ για την υπηρεσία μου και αυτό πιστεύω θα πρέπει να είναι το μέλλον. Έχει δίκιο επίση, δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή εγώ να σχολιάσω τα όσα πράττει η Βρετανική κυβέρνηση. Ελπίζω να συνειδητοποιεί ότι δεν θα πρέπει να χάσει την πάρα πολύ καλή φήμη που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ως ε, πρωτοπόρος βέλτιστων πρακτικών στην αστυνομική ε, δράση διεθνώς και επηρεάζουν πάρα πολύ ε, επηρέασαν στην εκπόνηση των νομοθετημάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πάρα πολύ καλή χέρι, πάρα πολύ καλή φήμη το Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει στο μέλλον να αυτό εξαιρεθεί. Και τέλος για το δουλεμπόριο, το trafficking το πρόβλημα στην αρχή ήταν εκτός Ευρώπης. Έφερναν γυναίκες και παιδιά για σεξουαλική εκμετάλλευση από την Ασία και την Αφρική, ενώ τώρα είναι κάτι που αφορά ένα πρόβλημα της Ένωσης της Σύριας. Πολλά από τα θύματα του τράφικινγκ είναι από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μιλούμε πια για Σέγγεν ή ελέγχου στα σύνορα. Δεν έχει πια σχέση αυτό με το πρόβλημα. Έχει Απόλυτο δίκαιο. Ε πρόεδρος. Παντού το βλέπουμε ε, στη γεωργία, στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, στην οικοδομή, στον κατασκευαστικό τομέα. Εργάζονται ε, ε, άνθρωποι σε πάρα πολύ επάνθρωπες συνθήκες και με πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς. Βεβαίως είναι γενικότερο το πρόβλημα και παγκόσμιο, γι' αυτό και έχουμε και πολύ καλές σχέσεις με όλους όπου συνεργαζόμαστε. Αλλά το πλαίσιο πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μοναδικό και μόνο στην Ευρώπη μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε την πιο ενοποιημένη και, ε, συνετή και συνεπή προσέγγιση. Θα ήθελα αυτό να το δω παγκοσμίω. Δεν γίνεται όμως με τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας βεβαιωθούμε ε, εμείς να συντονιστούμε, να συνεργαζόμαστε όσο γίνεται καλύτερα μεταξύ μας για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με τους άλλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Διευθυντά. Υπάρχουν δύο παρεμβάσεις. Ματιό πρώτα απ' όλα. Κυρία Ματιό, έχει το λόγο. Ένα ερώτημα. Αναφέρεται πολύ το ελευθερμπόριο τσιγαρών, ανθρωπίνων όντων, ε, παραποιημένα προϊόντα δεν μιλάμε ποτέ για το εμπόριο όπλων. Ε, τι γίνεται με τις καραμπίνες, με τα όπλα, μαχαίρια, τα καλάσνικοφ. Πού βρίσκεται η κατάσταση. Ε, κυκλοφορούν άτομα με όπλα και, και στη Μαρσαλία, στην πόλη μου, ε, έχουμε δει τέτοια γεγονότα. Υπάρχει όντως πραγματικά ε, παράνομο εμπόριο όπλων σε ποσότητες τώρα μιλάμε. Υπάρχει ένα εμπόριο όπλων που ξυπηρετεί εμπόλεμες καταστάσεις, το ξέρουμε αυτό, αλλά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουμε πόλεμο υπάρχει μια σημαντική, μίζωνος σημασίας δραστηριότητα εμπορίας όπλων είναι επικερδής αυτή η δραστηριότητα για τη μαφία. Θα είμαι επιγραμματική. Αναφερθήκατε σε ενδεχόμενε συνδέσει μεταξύ μαφία και τρομοκρατία. Υπάρχουν διασυνδέσει μεταξύ των διαφόρων μαφιόζικων οργανώσεων που είναι στι διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε. Και κάτι άλλο. Τι προσοχή δίδεται από εσά στις μαφίες. που βλάπτουν τους πάντες. Όσον αφορά τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες, που νομίζω ότι έδωσαν καλά αποτελέσματα, γιατί δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο, γιατί δεν αυξάνονται, νομίζω ότι είναι το εργαλείο εκείνο το οποίο θα πρέπει να είναι το χρησιμότερο για να μπορέσει να οδηγήσει στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών για τις έρευνες. Ένα λεπτό για τον κύριο Μακιντάρ, την κυρία Μάκιντάρ. Πολύ γρήγορα, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι ο κύριος Κέρκοπ αναφερόταν στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όχι του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου που είπε ότι δεν συνεργάζεται πλέον σε τόσο σημαντικά θέματα. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξής και αφορά περισσότερο την υποχθόνια αυτή η φύση, καταχθόνια φύση που λειτουργούν εν κρυπτό αυτοί. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες οργανώσεις, ο κ. Big που μπορούμε να στοχεύσουμε. Είναι σαν κάτι σαν μούχλα σε ένα κτίριο. Ε, άρα χρειάζεται διαφορετική ε, προσέγγιση για την καταπολέμηση. Έχετε κάποια παραδείγματα? Το πώς αλλάζει δηλαδή ο τρόπος καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας το δώσετε. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το εμπόριο όπλων είναι βασική δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος και χρειάζεται να χρησιμοποιούν τα όπλα για να επιβάλλουν τη δουλειά τους οι οργανώσεις αυτές. Μάλλον βλέπουμε τάση προς χρήση πιο επικινδύνων όπλων. Η κυρία Ματιέ αναφέρθηκε στα Καλάσνικοφ. Βλέπουμε όλο και περισσότερα στοιχεία να χρησιμοποιούνται Καλάσνικοφ περισσότερο παρά πιστόλια. Για να επιβάλλουν, να προστατεύσουν την επικράτειά της στο έδαφος τους έναντι άλλων εγκληματικών ομάδων. Να προστατεύσουν τον χώρο τους. Άρα υπάρχει επικίνδυνη τάση προς πλέον βαρέα επικίνδυνα όπλα σε πολλά μέρη της Δυτικής Ευρώπης και αυτό δημιουργεί αυξανόμενες ε, ανησυχίες για την ασφάλεια του κοινού, βέβαια. Είναι κληρονομιά των πολέμων στα Βαλκάνια πριν από 20 και 30 χρόνια. Πολλά παράνομα όπλα κυκλοφορούν σαν κληρονομιά των πολέμων. Πολλά τα συνδικάτα χρησιμοποιούν τους δικούς τους εμπόρους και προμηθευτές όπλων. Νέο φαινόμενο τα παράνομα αυτά όπλα ε, πολλούνται μέσω του διαδικτύου. Άρα online πολλούνται όπλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, παρέχονται όπλα μέσω του διαδικτύου. Τώρα συνεργασία μεταξύ κάποιων μαφιόζικων ομάδων σε διάφορες χώρες. Ναι, σίγουρα αυξάνεται η συνεργασία. Τα παραδοσιακά εθνικά όρια καταργούνται τουρκικές ομάδες, αλβανικές ομάδες, βρετανικές ομάδες κινούνται στην ίδια επιχείρηση, είναι εγκληματική και ο καθένας ασχολείται με παρανομή, ε, με προμήθεια διανομή ε, ενό παράνομου προϊόντος, άρα γίνεται κατανομή εργασίας μέσα στην παράνομη οικονομία ανάλογα με την εξειδίκευση κάθε παράνομης ομάδας. Και γίνονται όλο και πιο έξυπνοι και πιο επαγγελματίε από ό,τι και το παρελθόν. Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει στο βαθμό που συνεργάζεται, συνεργάζονται οι Ιταλικές οργανώσεις. Χρειάζεται στενότερη συνεργασία μεταξύ Europol και Ιταλικών αρχών στον τομέα. Μπορούμε να επιφέρουμε πολλές βελτιώσεις και θα ήθελα να εστιαστούμε εκεί. Να δούμε τι υποστήριξη μπορούμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη στο μέλλον. Δεν είδα το έγκλημα που εσείς αναφέρατε. Δεν είδα τέτοια σημάδια του οικονομικού παρεξήγησε αυτά που είπε ο κύριος ε, Κέρκοπ, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μαγνώ αυτό, αγνοείται αυτό που υπόθηκε. Όλα τα κράτη-μέλη όμως σίγουρα πρέπει να υποστηρίξουν την προσπάθεια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Συνεργασία να υποστηριχθεί. Θα μπορούσα να απαντήσω σε πολλά άλλα στοιχεία, ίσως κυρία Πρόεδρε, όμως θέλετε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πρόεδρος, Νέα, κύριε Διευθυντά, σα ευχαριστώ που δεχθήκατε να συζητήσουμε. Επαναλαμβάνω τι ευχαριστίες που δεχθήκατε την πρόσκλησή μας και θα έχουμε άλλες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και επαναλαμβάνω απευθυνών στους συναδέλφους ότι υπάρχει ανάγκη από την πλευρά μας κυρίως να χρησιμοποιήσουμε τη θεσιμότητά σας ούτω ώστε να εστερνιστούμε αυτά τις γνώσεις σας. Και σα ευχαριστούμε για την ευαισθησία που επιδεικνύεται έναντι των εργασιών μας. Εδώ ολοκληρώνουμε αυτό το πρώτο γύρο, το πρώτο τμήμα της συνεδριάσεώς μας. Με ανταλλαγή απόψεων τώρα με τον κύριο Ζων Φρανσουά Γκέιρου που είναι αστυνομικό διευθυντή ειδικού σώματο ε, υψίστου επίπεδου για έρευνες στη Γαλλία. Κύριε και πέρα ότι εκπροσωπείτε τι γαλλικές αρχές, είστε και εμπειρογνώμων στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματο. Θα ακολουθήσουμε την ίδια μέθοδο. Δίνω αμέσω το λόγο στον Φασουά Γκέιγο και μετά στου βουλευτέ. Έχετε το λόγο κύριε Γκέιγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι καλημέρα σας να επενθυμίσω ότι το πρωί, σήμερα το πρωί βρίσκομαι εδώ πέρα ε, και το κάνω αυτό ιδιωτικά θα έλεγα, όχι επίσημα από τη γαλλική πλευρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αντιμετωπίζει τέσσερις προκλήσεις ε, για το έγκλημα στρατηγικού επίπεδου. Καταρχήν θα πρέπει να αντιμετωπίσει δράσεις, μεγάλες εγκληματικές ε, δράσεις που ξεπερνούν τα εθνικά όρια, ενδογενείς, εξωγενείς. Ε, ορισμένες από αυτές τις δραστηριότητες είναι κλασικές ε, εγκληματικές δραστηριότητες, μαφία που λέμε, ε, μυστικές επιχειρήσεις. Αλλά αυτός εδώ, αυτή η δραστηριότητα της μαφίας έχει τέσσερις ιδιαιτερότητες. Η πρώτη έχει να κάνει με την πολλαπλή δράση, χωρίς κάποια εξειδίκευση, ευκαιριακά δηλαδή μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε όλες τις ευκαιρίες ε, όπως προκύπτουν. Μόλις δημιουργείται μια ευκαιρία, αυτές οι ομάδες ε, δράνε ή σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας ε, και διαδοχικά μπορούν να ασχοληθούν με θέματα προστασίας, ναρκωτικά, ε, παράνομα στοιχήματα. Δεν έχουν κάποια ιδιότητα, περνάνε από μια δραστηριότητα στην άλλη, όπου υπάρχει εκτίμηση κόστους όφλους. Δεν έχουμε δηλαδή ένα τομέα, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι θα λέγαμε κάνουν ε, δομημένα μια εγκληματική δραστηριότητα. Δεύτερη ιδιαιτερότητα. Αυτοί οι μεγάλοι οργανισμοί έχουν συχνά κάποια βάση, εδραιώνονται κάπου. Δημιουργούν ένα περιβάλλον το οποίο είναι ε, πρόσφορο για αυτές τις οργανώσεις. Ένας βιότοπος εγκληματικός θα λέγαμε αυτό έχει αποφασιστικό ρόλο, διότι δημιουργούν μια μεγάλη δύναμη. Αλλά δεν είναι μια παγιωμένη κατάσταση, επεκτείνεται. Έχουμε τις τέσσερις μαφίες στην Ιταλία, έχουμε τις φατρίες στις Αλβανόφωνες και την επέκτασή του στην Ευρώπη μέσα σε μερικές δεκαετίες. βλέπω το βραϊκό ε, επικράτεια η οποία έχει ε, οδηγηθεί σε μια ε, τέτοια κατάσταση. Το θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Επικράτητα πόσα θα λέγαμε κράτη μαφιόζικα περιέχει. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Τρίτη ιδιαιτερότητα. Αυτές οι οργανώσεις έχουν την ιδιότητα να προσαρμόζονται στις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές και απ' την άλλη δείχνουν μια ανθεκτικότητα στην καταστολή. Δεν καταφέρνουν τα κράτη να τις εξαλείψουν. Τέσταρτη ιδιαιτερότητα. Οι οργανώσεις αυτές ε, έχουν να κάνουν με οικονομική διακίνηση, μακροοικονομικά, που έχει μεγάλες επιδράσεις πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά. Πολλές φορές υπάρχουν οργανώσεις με ένα ΑΕΠ, θα λέγαμε, το οποίο να ξεπερνάει ορισμένες αυτό των μικρών χωρών. Βλέπουν δηλαδή ότι αποτελούν μεγάλες ε, σφαιρικές ε, δυνάμεις και δεν έχουν να κάνουν με μια δραστηριότητα περιθωριακή. Εδώ έχουν να κάνουμε εξουσία. Επίσης υπάρχει μια γεωγραφία όσον αφορά την κλιματικότητα στην Ευρώπη. από τη μια θα λέγαμε ότι έχουμε ένα είδος ένα μαφιόζικο τόξο από τη Μεσόγειο προς το Βορρά. Έχουμε τις ε, αλβανικοί μαφίες, τις αλβανόφενες και, τους, και την τουρκική, οι οποίες έχουν επεκταθεί σταδιακά προς το Βορρά. Γι' αυτό στο εγγύς μέλλον θα πρέπει να δούμε ότι υπάρχει η δημιουργία μιας γκρίζας ζώνης της είσοδο, θα λέμε, της Ευρώπης μια δεύτερη πρόκληση τώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει τι επιπτώσεις που θα υπάρχουν μακροοικονομικά. Τρει παρατηρήσεις. Πρώτη, η απορρίθμιση το, ε, στον, των εικονόγων αγορά ε, έχει οδηγήσει σε μια διευκόλυνση πούμε, όσον αφορά την ε, όρεξη αυτών των οργανώσεων. Οι φέρει φερρυπίν από, την, ε, ε, από τις επιπτώσεις στον φόρο για τον άνθρακα φερρυπίν οδήγησε σε, ένα, σε μια ζημία της τάξης των 1,5 δισεκατομμύρια για την, Ευρώπη, ε, για τη Γαλλία, 5-6 για την Ευρώπη. Επίσης, να αναφερθούμε τα προβλήματα που δημιουργούνται με τους φορολογικούς και τραπεζικούς παράδεισους και τα προβλήματα με τα μέσα που έχει κανείς σε επίπεδο δικαιοσύνης. Μια τρίτη παρατήρηση τέλος. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η τάση ας και στον χώρο, τον επίσημο χώρο των αγορών των δημοσιονομικών όπου έχουμε να κάνουμε πραγματικά με αρπακτικά. Έχουμε να κάνουμε μεγάλες ε, απάτες που γίνονται σε αυτό το χώρο και τα 30 χρόνια έχουν δημιουργηθεί απορριθμίσεις που έχουν οδηγήσει σε έγκλημα. Η φούσκα, η ακινήτων στη ΣΥΠΑ είχε τέτοιες επιπτώσεις και βλέπουμε ότι αυτοί που ήταν ακατεμένοι σε, αυτό, αυτή την υπόθεση παραμένουν σήμερα τιμόρυτοι. Τρίτη πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει ένα κυβερνοχώρο ο οποίος θα λέγαμε είναι ένας χώρος ανομίας. Είναι ένας χώρος ευάλωτος στην εγκληματική δραστηριότητα και έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Ξεπερνάει τα εθνικά χώρα, ε, όρια και είναι ρευστός βλέπουμε σε αυτόν τον χώρο, τον ε, εικονικό, ε, υπάρχει μια μεγάλη κίνηση, κινητικότητα μάλλον. Φερρυπίν, στο, στο χώρο το, το, του αθλητισμού υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι πόροι, διακίνηση χρημάτων και εκεί πέρα έχουμε Φερρυπίν την εγκληματικότητα που έχει να κάνει με τα σημαίνα παιχνίδια. Και αυτό γίνεται σε όλη ε, την παγκόσμια θα λέγαμε επικράτεια. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει υπόψη και τις συνέπειες της οικονομικής και διεθνική κρίσης που έχει να κάνει με την ε, φούσκα στα ακίνητα στην Αμερική. Ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία, ιστορική θα λέγαμε, για το, ε, οργανωμένο έγκλημα. Και υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, τα κράτη ε, τα οποία έχουν προβλήματα σε επίπεδο προπολογισμών έχουν κάνει μειώσει όσον αφορά στο αστυνομικό ε, χώρος, στα θελωνία, στην δικαιοσύνη. Επιπίσεις έχουν να κάνουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ε, κεφάλαια με νόμιμο τρόπο μέσω του τραπεζικού συστήματος. Συχνά πολλές τέτοιες επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρές που πάνε πηγαίνουν σε αυτό που λέμε shadow banking που ελέγχεται από το οργανωμένο έγκλημα. Και με αυτόν τον τρόπο αυτός ο χώρος που έχει μεγάλες δυνατότητες διεισδύει στην νόμιμη οικονομία. Οι συνέπειες αυτών των φαινομένων δεν, ναι, είναι αθέατες θα λέγαμε, αλλά έχουν βάθος και διάρκεια. Επίσης να δούμε τη μεγάλη διαφορά όσον αφορά τη δραστηριότητα των τρομοκρατών. Η τρομοκρατία είναι ορατή με πιο περιορισμένη ε, αρνητική επίπτωση, αλλά το οργανωμένο έγκλημα είναι αθέατο, αλλά έχει μεγαλύτερε επιπτώσεις. Ξέρουμε πολύ καλά ότι στην κοινωνία της πληροφόρησης και ενημέρωσης κάτι το οποίο δεν περνάει στα ΜΜΕ μπορεί να έχει μια διάρκεια και να επιβιώσει ατιμωρητή. Υπάρχει συστηματική διαφθορά και μπορούμε να μιλάμε για την δημιουργία μιας εγκληματικής μπουρζουαζίας. Έχουμε περάσει δηλαδή από το αόρατο χέρι στο εγκληματικό χέρι που ελέγχει τα πράγματα. Ελέγχουν ε, λίγο πολύ τέτοιες καταστάσεις που οδηγούν σε συνέπειες και στους προπολογισμούς των χωρών ε, μελών. Στην υγεία, στο περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε ότι το οργανωμένο έγκλημα μεταλλάσσεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο και διασυνδέεται με δύο τομείς. Απ' τη μια την τρομοκρατία και απ' την άλλη με αυτό που λέμε η εγκληματικότητα των χαρτογιακάδων. Εμείς πρέπει να δείξουμε ετοιμότητα για αυτές τις ε, αλλαγές στο συγκεκριμένο πλαίσιο σήμερα, διότι είναι το κατάλληλο για την ε, επέκταση αυτού του συστήματος. Υπάρχουν ε, ε, κάποιοι παράγοντες στους οποίους πρέπει να θίξουμε όσον αφορά τις επιπτώσεις μακροοικονομικά. Καταρχήν έχουμε την βαλκανοποίηση, τον καταγερματισμό του κόσμου. Από το 45, από περίπου 40 χρόνια, περάσαμε σήμερα στην ύπαρξη 200 κρατών, τα οποία θα λέγαμε είναι χώρες ποτέμκιν, ε, ευάλωτα, αδύναμα. Μετά έχουμε την παγκοσμίεση, ε, όπως είναι γνωστό να λέγεται. Τέλος, τη γενικότερη εμπεραματοποίηση Τέταρτον, την απορρίθμιση, τη δογματική απορρίθμιση των αγορών. Αυτή δημιουργεί εγκληματικότητα. Δίνει ευκαιρίε για δραστηριότητε εγκληματικέ μεγάλη έκταση. Μετά έχουμε τι επιπτώσει από τον αγώνα κατά τη τρομοκρατία. Και τέλο, οι συνέπειε ε, της τη χρηματοπιστωτική κρίση. Συμπερασματικά, στον χαοτικό κόσμο που έχουμε μετά το ψυχρό πόλεμο, το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μια μεγάλη στρατηγική πρόκληση που ξεπερνάει τα θέματα που έχουν να κάνουν με δικαιοσία και όργανα καταστολής. Για να υπάρχει επιτυχία σε αυτόν τον αγώνα χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, μια συνεχή εργασία γνώσης, παιδαγωγίας και να ξεφύγει κανείς από την και να μην εθελοτοφλούμε. Δεν μπορεί να πολεμήσει κάτι το οποίο κανείς αγνοεί, αρνείται ή δεν παίρνει στα σοβαρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια τέτοια επιτροπή ε, κοινοβουλευτική, διότι ε, μπορεί να ενημερώσει και να επηρεάσει αυτούς που παίρνουν αποφάσεις. Και τέλος, να δώσουμε μια προτεραιότητα στην κατάρτιση. Να γίνει δηλαδή μια δουλειά μεθοδικά, ε, με σωστό τρόπο και δράσεις οι οποίες να προλαβαίνουν. Όχι... Ευχαριστώ κύριε Γκέιρο για την ε, ακρίβεια με την οποία κάνατε την παρουσίασή σας. Ε, μπορούμε να δώσουμε αμέσω το λόγο στις ομάδες ξεκινώντας ε, με τον κυρία Ματιέ του ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση που έκανα και δεν είχα απάντηση αυτήν, θα την ξαναθέσω. Τι λέτε, είναι ένα θέμα εξουσίας, είναι ένα φαινόμενο αυτό του οργανωμένου εγκλήματος ή έχει να κάνει μόνο με οικονομική διάσταση. Εσείς πρέπει να ξέρετε. Δεν μπόρεσε κανείς ποτέ να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα διότι η... Ε, αυτό που έχει απέναντι σε αυτές άσχετο από ποια χώρα είναι, πάντοτε δεν πετυχαίνει το στόχο του. Τι γίνεται, θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί με μια νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι να περιοριζόμαστε σε μέσα από είναι εθνικής ε, φύσεως. Ευχαριστώ. Σκοτσέτα έχει το λόγο. Για το ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πραγματικά για την ανάλυση που κάνατε, που ήταν σύντομη μεν, αλλά λεπτομερέστατη δε. Διότι κάθε σημείο που θίξατε χρειάζεται ώρες εμβάθυνσης. Ήσασταν αποτελεσματικότατος και θέσατε το πλαίσιο. Θέσατε το πλαίσιο, πιστεύετε, του οργανωμένου εγκλήματος που εδράζεται επί της παραδοσιακής αναλύσεως που κάναμε για τη μαφία. Για την Κόζα Νόστρα περισσότερο από ότι για τη μαφία. Το μοντέλο Κόζα Νόστρα ελέγχει την επικράτεια και οι ομάδες που παρουσιάζονται στην Ευρώπη με συνδετικό τρόπο ελέγχουν την επικράτειά τους. Το στόχο αυτό ότι γίνονται στοιχεία αστικά ποινικού τύπου. Μια μπουρζουαζία. Και θέσατε και το θέμα και τις ασπίδες που θέτουν σε επιχειρήσεις τους κάνουν νόμιμες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν νόμιμα συστήματα αυτές, αυτή ε, η ε, μαφιόζικη μπουρζουαζία. Άρα σχετίζεται παράνομη δραστηριότητα με νόμιμη δραστηριότητα και το θέμα με τις παρεκκλήσεις πολιτικές που αναφέρατε. Την ανάλυση τη συμμερίζομαι που κάνατε. Ε, εδώ και χρόνια μερικοί από εμά το βλέπαμε έτσι το θέμα ήταν κάτι κατεπήγον κατά το παρελθόν και τώρα έχει γίνει κάτι μόνιμο στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρώπη, σαν φαινόμενο. Πρέπει να βρούμε αντίδοτο. Βλέπω δισταγμού παράξενου σήμερα στην Ευρώπη. Το συζητούμε, τα διάφορα ποινικά συστήματα των κρατών μελών είναι πρόβλημα και τίθεται συνέχεια τα ίδια ζητήματα. Πρέπει να έχουμε κοινά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτά που αναφέρθηκαν. Προέρχομαι από, από γη της μαφίας και συμμερίζομαι αυτά που υπόθηκαν και είδα τι αλλαγέ τη μαφίας. Είπατε ότι το οργανωμένο έγκλημα ε, συνδέεται περισσότερο με τις υποθέσεις και με την εγκληματική μπουρζουαζία που κινείται σε επιχειρήσεις, όχι τόσο πολύ με τα προβλήματα τα οικονομικά. Α, σαν πολιτικό σύστημα, σαν χώρε πρέπει να το συμμεριστούμε αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε οδηγίες κοινέ που να μην δημιουργούν κενά και να είναι στοχευμένες. Τι θα προτείνατε σαν νομοθεσία εσείς για αποτελεσματική καταπολέμηση αυτού του είδους των οργανωμένων ομάδων, του οργανωμένου εγκλήματος, εγκλήματος που μεταμορφώνονται οι ομάδες ε, και που γίνονται πολύ δύσκολα αντιμετωπιστούν από εκείνους που δεν έχουν ε, εμπειρία για αυτό το, όσον αυτό το θέμα. Ευχαριστώ από πλευρά για δύο λεπτά. Ο κύριο Νιούτον Ντόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, εδώ είμαι. Είπατε βαλκανοποίηση του κόσμου. Αυτό είναι το βασικό που ξεχώρισε αυτά που είπατε. Αν σας δίναμε εξουσίες, ποιο είναι το όραμά σας. Πώς θα καταπολεμήσει ο κόσμος και η Ευρώπη τη βαλκανοποίηση των εθνικών εξουσιών και τη δυνατότητα καταπολεμήσεως του εγκλήματο σε παγκόσμια κλίμακα. Τι θα κάνατε εσείς. Αυτή είναι η ερώτηση. Γκουε, ο κύριος Σόντεργκάρτ για ένα δίλεπτο. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτά που μας είπατε. Έχω μία δύο να σας θέσω. Συνεργάζεστε από ό,τι κατάλαβα με τον όρο του χρεοκοπημένου κράτους, όπως και στην δημοκρατία, failed state. Αλλά λόγω της βαλκανοποίησης που επίσης αναφέρατε, Αυτέ οι χρεοποιημένε χώρε, οι αποτυχημένε χώρε μπορεί να χρησιμοποιηθούν από παράνομε ομάδε, από ό,τι κατάλαβα. Μπορείτε να μα δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε όσον αφορά την χρήση των failed states από τι εγκληματικέ οργανώσει. Και για τι χρηματοπιστωτικέ αγορέ, τι ε, απορριθμισμένε, πόσο ενίσχυσαν αυτέ τι ε, εγκληματικέ συμμορίε. Τι μηχανισμούς βλέπετε που χρησιμοποιούν και λειτουργούν. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για τον κύριο Γιακολίνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Άκουσα και εγώ με τα ζωηρού ενδιαφέροντος την παρέμβαση που μόλις έλαβε χώρα. Από την οποία διεφάνει σαφέστατα ότι το εγκληματικό φαινόμενο είναι ένα φαινόμενο που έχει σχέση με την επικράτεια δαφική και με την πολιτική. Και είναι προφανής οι διασυνδέσεις. Πρέπει να βρούμε και πολιτικές ε, λύσεις αν θέλουμε νομοθετικές. Άρα θέλαμε να δούμε ποιες σκέψεις έχετε σχετικά με το νομοθετικό πανόραμα που έχουν δημιουργήσει τα διάφορα κράτη-μέλη και που διαφέρει από χώρα σε χώρα. Έχουμε επαρκή επίγνωση αυτού. και πόσο σημαντική είναι η παρουσία των κλιματικών οργανώσεων και κυρίως εκεί που το έπινε κάτω από τα πρότυπα, κάτω από το μέσο τον ευρωπαϊκό. διότι δυσδύει η μαφία ιδιαίτερα στις περιοχές όπου δίδονται και πολλά χρήματα από τα ιδιωτικά ταμεία και υπάρχει υποστήριξη. Θέλω τη σκέψη σας πάνω σε αυτό η έκθεση πρέπει να έχει ένα σημείο αναφορά, όχι μόνο για του άλλου φορεί τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά πρέπει να δώσουμε και κάποια κίνητρα για το πλησίασμα εναρμόνιση των διαφόρων νομοθεσιών που εμποδίζει κάπως την εργασία την αστυνομική και τη δικαστική ούτως ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η μαφία και αυτού του συγκληματικές οργανώσεις. Ευχαριστώ κύριε Γιακολίνο. Ο κύριος Μίσκη έχει το λόγο για ένα λεπτό. Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Θα ήθελα να προσθέσω ότι είχαμε πολύ ενημέρωση στατιστικά στοιχεία. Παρ' όλα αυτά δεν έχω καταλάβει πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Ίσως θα πρέπει να θυμόμαστε ποιος είναι ο βασικός στόχος των εγκληματιών. Το χρήμα αν ένας κακοποιός έχει δυσκολίες στη πρόσβαση και στη χρήση του χρήματος, τότε θα έχουμε πετύχει να μειώσουμε τα επίπεδα του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πάρουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για τον κύριο Σμιτ, τελευταία παρέμβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Μπορεί να σας πω ότι θεωρώ ότι η απορρίθμιση στην ε, ε, αγορά, στην οικονομία δεν είναι το πρόβλημα. Μπορεί να είναι ένα πρόβλημα, αλλά αν καταφέρουμε να κλείσουμε τα παραθυράκια ε, στη ρύθμιση της αγοράς, τι θα γίνει, θα εξαφανιστεί το οργανωμένο έγκλημα, δεν πιστεύω. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να εγκληματεί κανείς. ακόμα και αν οι χρηματαγορές δεν είναι απορριθμισμένες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κογκρέσο αποφάσισε να γίνει αυτή η φούσκα ε, στην κτήματα αγορά στι Ηνωμένες Πολιτείες που έσκασε τελικά. Εγώ ήμουν στην Επιτροπή για την κρίση και είχαμε διάφορους λόγους εντοπίσει, αν δεν απατώ με 38, για τη χρηματοπιστωτική κρίση. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι παρόδο. Ερώτηση τώρα. Χρειαζόμαστε πραγματική ομοσπονδιακή ε, αστυνομία στην Ευρώπη όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό θα μας βοηθήσει για να καταπολεμήσουμε το έγκλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, πριν σας δώσω το λόγο, να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για την έξοχη σύνοψη παρουσιάσατε και την ικανότητα με την οποία παρουσιάσατε τόσο σύντομα μέσω ενός πλαισίου πληρέστατου όχι μόνο τα προβλήματα, αλλά και τις ενδεχόμενες λύσεις που πρέπει να δοθούν από τα θεσμικά όργανα. Ερώτηση. Από την εμπειρία σας, χρειάζεται ομοσπονδιακή αστυνομία αυτό που έθεσε ο κύριος Σμιτ. Εγώ ρωτάω όμως, από τη δική σας άποψη, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ενιαίο νομοθετικό, ένα μοναδικό νομοθετικό κείμενο κατά το οργανωμένο εγκλήματος. Ο κ. Μπορσελίνο είπε ότι θα έπρεπε να Υπάρχει ένα 416α ευρωπαϊκό. Να αναγνωριστεί λοιπόν το αδίκημα αυτό του συνεταιρίζεσαι για σκοπούς τέτοιου, της δημιουργία ομάδας για τέτοιου παράνομους σκοπούς. Να θεωρείται αδίκημα, έγκλημα. Θεωρείται λοιπόν ότι χρειάζεται μια τέτοια ενοποίηση των διαφόρων ποινικών συστημάτων τη ποινική νομοθεσία. Θα κοιτάξω σύντομα να απαντήσω σε όλες αυτές τις παρατηρήσεις, υπενθυμίζοντας ε, ξανά ότι, ότι δεν εκπροσωπώ επίσημα κάποια αρχή της Γαλλίας. Καταρχήν, στην πρώτη ερώτηση που μου έγινε, ναι, τα φαινόμενα ε, της εγκληματικής δράσης σήμερα είναι φαινόμενα τα οποία δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε τάση προς εξουσία. Υπάρχουν δηλαδή αυτές τις δραστηριότητες στη, με τη μαφία Φερπίν στην Ιταλία. Ξεκινάει σε φατριακό επίπεδο, έχει όμως πρόσωπο προς τα έξω έχει δραστηριότητες με επιχειρήσεις ε, καταχωρημένες νομικά υπάρχουν δηλαδή όλες οι πτυχές, οι πολιτικές, οι οικονομικές, κοινωνικές και έχουν ένα ρόλο ο οποίος δεν είναι περιθωριακός. Και κάτι τέτοιο μπορούμε να δούμε και σε άλλα μέρη της Ευρώπης με άλλη μορφή οργάνωση. πάρα πολλές φορές θέχτηκε το θέμα τι, θα κάνει η Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το θέμα δηλαδή μιας να έχουμε ε, καθορισμένα επίπεδα στο νομικά μέσα που έχουμε για να μπορέσουμε να κάνουμε συντονισμένες ενέργειες. Ε, παράλληλα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, οι χώρες ε, δεν μπορούν να αποποιηθούν τις ευθύνες τις εθνικές που έχουν. Ε, δεν μπορούν δηλαδή οι χώρες να, να μην κάνουν, ε, να αποφύγουν να κάνουν κάποια πράγματα θεωρώντας ότι υπάρχει από πάνω κάτι το οποίο είναι ευρωπαϊκού επίπεδου και ξεπερνάει τα, τα κράτη-μέλη. Κανένα, καμιά χώρα δεν θα μπορούσε να κάνει για λογαριασμό των Ιταλών αυτό πρέπει να κάνουν οι ίδιοι, το ίδιο ισχύει για τη χώρα μου και για όλες τις άλλες. Ε, λοιπόν, η πρώτη ευθύνη είναι η ευθύνη των κρατών. Τώρα, ακόμα και να εξασφαλίσουμε μια, ε, ένα δικαστικό ε, επίπεδο το οποίο είναι εναρμονισμένο, θα υπάρξει κάποια προβλήματα. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που έχουν καλύτερα συστήματα, τα οποία όμως δεν εφαρμόζονται είτε γιατί δεν υπάρχει η βούληση, είτε δεν υπάρχουν τα μέσα. Το Μεξικό σίγουρα έχει την καλύτερη νομοθετική, ας πούμε, ε, ε, τις καλύτερες νομοθετικές ρυθμίσεις για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ε, εμπόρους ναρκωτικών. Για τη βαλκανοποίηση του κόσμου που ανέφερα. ο κόσμος έχει εξελιχθεί. Αναφέρθηκαμε 45 κράτη που πήγαν το τέλη του 40, τώρα έχουμε 200. Μπορεί στις επόμενες δεκαετίες να έχουμε και 10-20 επιπλέον κράτη. Αυτό είναι ένα ιστορικό φαινόμενο. Είχαμε την ε, διάλυση των ε, κρατών που είχαν ε, τις απικίες Υπάρχουν όλες ε, οι διάφορες αιτίες που οδηγήσαν σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και για αυτό το πράγμα και ούτε χρειάζεται να, να αξιολογήσουμε να... αυτό το φαινόμενο. Το θέμα είναι οι συνέπειες. Πολλά από αυτά τα νέα κράτη πραγματικά δεν έχουν ε, δυνατή υποδομή ε, θεσμικά όργανα, αστυνομία, δικαστικό σώμα για να μπορέσουν ε, τελωνία για να αντιμετωπίσουν τα πρόβληματα. Και σε αυτές τις χώρες ε, ο συσχετισμός δυνάμεως είναι αντίθετος. Βλέπουμε δηλαδή σε, αυτές, σε ορισμένες από αυτές τις χώρες έχει ανατραπεί ο συσχετισμός δυνάμεως όπως είπα και παίρνουν το πάνω χέρι αυτοί που είναι στο περιθώ... κατά τα άλλα στο περιθώριο εγκληματικέ οργανώσεις. Δεν θα επανέλθω στο θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα subprime και με την απορρίθμιση των αγορών. Δεν θα με κάνετε να, να αποφύγω την ιδέα ότι ε, το θέμα αυτό είχε να κάνει με συστημική απάτη η αγορά κινήτων στην Αμερική. Και θα τελειώσω εκεί που ξεκίνησα. Ότι είναι σημαντικό και να υπάρξει μια ε, ξεκαθορισμός ε, κοινών ε, ε, μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν κάποια ευαισθησία. Έχουμε την ιστορία ε, του οργανωμένου κλίματος, η μαφία, αλλά επιμένω χρειάζεται να ενημερωθούμε, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε. Δίνω μεγάλη έμφαση σε αυτό το θέμα της γνώσης. Το οργανωμένο κλίμα είναι περίπλογο. Καταφέρουν να εγκατασταθούν σε ένα χώρο και να διεισδύσουν στο οικονομικό και πολιτικό ιστό. Σας ευχαριστώ κύριε Γκέγου. Πάνω απ' όλα για το πάθος με το οποίο μας μιλήσατε και για το χρόνο που μας διαθέσατε. Δεν είναι απλό να βρει κανείς έναν μη Ιταλό διότι εμείς είμαστε από τη γη της μαφίας, που να κάνει ένα τέτοιο, μια τέτοια ανάλυση και που διαπιστώνει αυτές τις ανάγκες. Ευχαριστώ εκ καρδίας, εξ ονόματι όλης της Επιτροπής που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Σας ζητώ ή δυνατόν να μας δώσετε ένα αντίγραφο της ομιλίας σας. Α, την έχουμε ήδη. Σας ευχαριστώ. Θα διανύμουμε το κείμενο. Ευχαριστώ. Με την παρέμβαση λοιπόν του κυρία Γκέιγο τελειώσαμε το πρώτο θέμα, προβληματισμό επί του πρώτου θέματος, με την παρέμβαση του Αντιπροέδρου Κάλλος Ζάιν θα ανοίξουμε το παράθυρό μας προς το δεύτερο γύρο. Το δεύτερο θέμα θα συζητήσουμε. Ξεκινήσουμε την πρόεδρο Τζέιν και μετά θα συνεχίσουμε το απόγευμα. Χάρη στην παρουσίαση του πρόεδρου του Eurojust, Κάρλο Σέιερ, θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη συνεργασία και σύμπραξη μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς, το ξέπλυμα χρήματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σήμερα επανειλημμένα αναφερθήκαμε στη συνεργασία, στη σύμπραξη. Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε, μπορείτε να μας πείτε τι είναι η τρόπο μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε αυτές τις συνέργειες. Έχετε το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιτρέψτε μου καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που απευθύνατε στη Eurojust για να συμμετάσχει σε αυτή τη διακεκριμένη ομίγυρη. Ε, ζητώ συγγνώμη εξ ονόματος ε, της κυρίας Μισελ Κόνιγκς που είναι η πρόεδρος του Eurojust που δυστυχώς κολλείεται και δεν μπορεί να έρθει στη Βρυξέλλες σήμερα. Έχει άλλη ενηρημένη υποχρέωση γιατί συνεδριάζει η Ολομέλεια των Εθνικών Μελών της Eurojust και επίσης ε, έχει και μια παρέμβαση ε, να κάνει την Πέμπτη στην Επιτροπή Ελευθεριών όπου θα παρευρεθεί και ε, θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεση της Eurojust για το 2011. Σήμερα το πρωί άκουσα εγώ δύο πράγματα. Πρώτον ότι δεν λειτουργεί η Eurojust και το δεύτερο που άκουσα είναι ότι δεν λειτουργεί αρκετά καλά. Δηλαδή μεγάλη πρόκληση τώρα ε, μπροστά μου έχω για να σας πείσω ε, περί του αντιθέτου. Αλλά πιστέψτε μου, δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Η δική μου παρουσίαση έχει ως στόχο επίσης ε, ζητήματα που η συνεργασία και η λειτουργία της Eurojust μπορεί να βελτιωθεί. Και αν μου επιτρέπει ο χρόνος, μπορώ και να σας παρουσιάσω σύντομα ε, ένα περιστατικό, μια περίπτωση και να σας εξηγήσω με το παρόν ε, νομικό πλαίσιο ποιες ε, είναι οι δυσκολίες και οι περιορισμοί για τη Eurojust. Έχω επίγνωση του γεγονότος ότι μπορεί ακόμα να μην αναγνωρίζεται, να μην έχουμε ένα σήμα αναγνωρίσιμο στη Eurojust τύπου Coca-Cola, αλλά ε, να σας εξηγήσω λίγο την αποστολή, τα καθήκοντα της Eurojust, ε, τα μέσα και τους στόχους που έχουμε στη διάθεσή μας, και τα εργαλεία καλύτερα. Στη συνέχεια την απόφαση Eurojust το 2009 και τα μέσα που μας έδωσε για τη δουλειά μας ε, μετά θα αναφερθώ στο οργανωμένο έγκλημα, στη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος από τη σκοπιά της Eurojust και τέλος θα σας ε, δώσω και μερικά στοιχεία αριθμητικά και ενδεχομένω και δύο παραδείγματα για να σας ε, περιγράψω την κατάσταση. Ερχόμενος τώρα στο νομικό πλαίσιο, να θυμίσω ότι δημιουργήθηκε το 2002 Eurojust μετακόμισε στη Χάγη τέλη του 2002 επίσης και ε, η νέα απόφαση για τη Eurojust που ελήφθη το Δεκέμβριο του 2008 αλλά τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2009 ε, ορίζει τη σημερινή λειτουργία και έχει δώσει περισσότερες εξουσίες και αρμοδιότητες ε, στον οργανισμό στην καθημερινή του δουλειά. Γιατί τα λέω όλα αυτά και αναφέρομαι στη νέα απόφαση για τη Eurojust. Διότι κυρίως όλα τα κράτη-μέλη δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει αυτή την απόφαση και έπρεπε να την είχαν εφαρμόσει μέχρι τον Μάιο του 2011. Και στην καθημερινή μας δουλειά αυτό είναι εμπόδιο. Γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε ενδεχομένω πραγματικές χειροπιαστές επιτυχίες. Αλλά το νομικό πλαίσιο δεν είναι μόνο κάτι που ε, θεωρείται δεδομένο αλλά είναι κάτι το εξελισσόμενο. Να σας θυμίσω ότι δύο άρθρα της Συνθήκης Λισαβόνος ασχολούνται με το έργο της Eurojust ή αναφέρεται σε αυτές. Είναι το άρθρο 85 το πρώτο που αφορά τη δομή της εξουσίες και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της Eurojust όταν ε, μιλώ για κοινοβουλευτικό έλεγχο ε, αφορά αυτό την αξιολόγηση και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Επανέρχομαι στο άρθρο 85 λοιπόν. Να σας πω ότι βεβαίως η δομή της Eurojust μπορεί να βελτιωθεί και να είναι ακόμα πιο αποτελεσματική, αλλά κατά την άποψή μου, και όπως και κατά την άποψη του οργανισμού, υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο στο άρθρο 85, δηλαδή οι εξουσίες που μας εκχωρούνται είναι σημαντικές. Στο άρθρο 85 ας πούμε προβλέπεται δυνατότητα ε, έναρξης ερευνών ή πρότασης ε, και δίωξης. Θυμίζω την αποστολή της Eurosat σύμφωνα με το άρθρο 85 της Συνθήκης Λισαβόνας όπως βλέπετε στη διαφάνεια και έρχομαι ε, στο πραγματικό στόχο και σκοπό της μονάδας μας η απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου του 2000 του Συμβουλίου Εσωτερικών και Δικαιοσύνης όριζε ότι η αποστολή μας είναι να αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά και έρχομαι τώρα και στο πεδίο εφαρμογή και της δικής σας ε, επιτροπής ιδιαίτερα ε, πιο αποτελεσματικά σοβαρό διασυνοριακό έγκλημα ιδιαίτερα όταν είναι οργανωμένο και αφορά δύο περισσότερα κράτη-μέλη. Στόχοι της Eurojust είναι να ενισχύουν και να βελτιώνουν το συντονισμό των ερευνών και των διώξεων, να βελτιώνει τη συνεργασία με ε, αμοιβαία νομική συνδρομή και ε, έκδοση, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ένταλμα ε, Έκδοσης και υποστήριξη των αρμοδίων αρχών όταν πρόκειται για τη δίωξη διασυνοριακού εγκλήματος. Έρχομαι στα καθήκοντα της Eurojust, όπως προβλέπονται στα άρθρα 6 σε ό,τι αφορά τα εθνικά μέλη και το άρθρο 7 σε ό,τι αφορά ε, το συλλογικό σώμα, το κολέγιο ή την ε, ολομέλεια των εθνικών μελών. Ε, βασικός στόχος είναι να ερευνούν ή να ζητούν από τις απαραίτητες, τις αρμόδιες συγγνώμη αρχές να διώκουν ή να κάνουν έρευνες, να συνεργάζονται, να συστήνουν τινούν κοινέ ομάδες ερεύνης και το σημαντικό να ε, γίνεται ανταλλαγή απόψεων και ε, πληροφοριών. Έρχομαι τώρα σε ένα κρίσιμο σημείο του έργου μας. Προς το παρόν η Eurojust έχει μόνο την εξουσία να ζητάει πράγματα. Δεν έχει καμία εξουσία ή καμία δυνατότητα να επιβάλλει ή να υποχρεώνει ε, ε, σε μια δικαστική αρχή να προχωρήσει στην άσκηση ποινική δίωξης ε, σε άλλες έρευνες. Αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 85 της Συνθήκης Λισαβόνας, θα μπορούσε να ισχύει. Δεν θα επιμείνω στα υπόλοιπα καθήκοντα. Η Eurojust, εκτός από την επιχειρησιακή δουλειά της, στο λεγόμενο τρίτο επίπεδο που είναι οι συνεδριάση συντονισμού ε, έχουν σχέση ας πούμε με τη ε, διοργάνωση ταυτόχρονα σε διάφορα κράτη-μέλη συλλήψεων ή ε, ερευνών. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν σε μια συνεδρίαση συντονισμού στη Eurojust αλλά έχουμε και τεχνικές και στρατηγικές συνεδριάσεις όταν πρόκειται για ειδικέ ομάδες εγκλήματος ή, ε, ή ε, φαινόμενα. Και στο οργανωμένο έγκλημα. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω τα εξή τρία ζητήματα που εισάγονται από τη νέα απόφαση για τη Eurojust, η οποία νέα απόφαση ακόμα δεν εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη, θυμίζω, και σε αρκετά. Ε, το 1 τρίτο περίπου των κρατών μελών δεν εφαρμόζουν αυτή την απόφαση του 2009. Έτσι συμμετέχουμε λοιπόν σε κοινέ ερευνητικέ ομάδες. Ε, έχουμε την ε, λεγόμενη συνεργασία και συντονισμό on-call ε, και για ανταλλαγή ε, πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 13. Ε, οι ομάδες, κοινέ αυτές οι ερευνητικές ομάδες, είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία μας στο μέλλον και ενδεχομένω και σε άλλα θεσμικά όργανα θα χρειαστεί να συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο Γνωρίζετε ότι αυτές οι μικτές ερευνητικέ ομάδες στην αρχή ε, θεωρούν το κάτι το θνησιγενές. Δεν δημιουργήθηκαν στην αρχή πολλές τέτοιες ομάδες και ένας από τους λόγους πάντα ήταν η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης αυτών των ε, ομάδων. Μετά λήφθη μια πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εξασφάλισε τη χρηματοδότηση για αυτές τις ομάδες και 95% των κονδυλίων προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η Eurojust έδινε το υπόλοιπο 5%. Και μπορεί κανείς να πει πραγματικά ότι αυτή η χρηματοδότηση, η εξασφάλιση της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε μια σημαντική όθηση στη σύσταση αυτών των ομάδων. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω ότι η Eurojust το 2010 ή από το 2010 μέχρι και φέτος, τον Ιούνιο, υποστήριξε οικονομικά 65 μικτές ε, ομάδες έρευνας σε όλη την Ευρώπη. Επίσης, η απόφαση για τη Eurojust ε, ε, οδήγησε σε ένα συντονισμό on-call. Τι θα πει αυτό? Ότι είναι στη διάθεση ε, των διοκτικών αρχών και των ερευνητικών αρχών 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Για να σας δώσω ένα σύντομο ε, παράδειγμα ε, των εκτιμάτων αυτού του συντονισμού on call, σε επιφυλακή δηλαδή, πέρσι το Δεκέμβριο γύρω στις 10 το βράδυ μια μέρα με πήρε τηλέφωνο ένας Γάλλος συνάδελφος και μου είπε ότι οι γαλλικές αρχές εξετάζουν έναν ύποπτο ε, σε μια υπόθεση διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και ομολόγησε ότι είχε 3 εκατομμύρια ευρώ ο ύποπτος ε, σε ένα τραπεζικό λογαριασμό στο Λουξεμβούργο. Και επειδή ήταν εγκληματική οργάνωση, οι υπόλοιποι ε, δεν ξέραμε αν είχαν εξουεδότηση και πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό και καταφέραμε λοιπόν τουλάχιστον να παγώσουμε τα κονδύλια αυτά μέσα στη νύχτα, από τη μια μέρα στην άλλη. Σας είπα στις 10 το βράδυ με πήρε τηλέφωνο αμέσως ήρθα ε, σε επαφή με την αντίστοιχη υπηρεσία πληροφοριών, οικονομικών πληροφοριών του Λουξεμβούργου και στις 9 ε, το πρωί πριν ε, ανοίξουν οι τράπεζες είχε παγώσει ο λογαριασμός αυτός και στη συνέχεια κατασχέθηκε και επίσημα την ίδια μέρα. Είμαι πεπισμένος ότι εάν δεν είχαμε αυτό το συντονισμό, το τηλεφωνικό, το μόνιμο, δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα προς λοιπόν αυτή η ανταλλαγή προφοριών για να βελτιώνεται η δουλειά μας και στα κράτη-μέλη. Χρειάζεται οπωσδήποτε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τη νέα απόφαση για τη Eurojust. Επίσης, ε, θα ήθελα να θυμίσω τη συνεργασία μας με τη Europol. Θα βρείτε ε, τις λεπτομέρειες ε, στη διαφάνεια που βλέπετε από πλευράς πρακτικής λειτουργίας και καθημερινής δουλειάς. Επιμένω ότι η Eurojust θα πρέπει να συνεργάζεται με την Europol σε βασικά σημεία. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με 17 focal points, αλλά η Europol δημιουργήθηκε κυρίως για αναλυτικούς σκοπούς, ενώ η Eurojust κυρίως για επιχειρησιακούς σκοπούς. Για μας ε, είναι λογικό, τουλάχιστον έτσι μας φαίνεται, να συμμετέχει η Eurojust σε όλες τις ε, δραστηριότητες στα focal points της Europol, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας. Ε, η πρώην AWF, analysis ε, work files, Hydra και Dolphin. Hydra και Τώρα έχει μπει σε μια ταχύτητα πορείας σε υπόθεση αυτή και ε, το 2011 η Όλαφ ε, παρέπεψε στη Eurojust 8 περιπτώσεις και ε, ήταν παρούσα σε 8 συνεδριάσεις συντονισμού. Εδώ θα δείτε πέρυσι ότι αντιμετωπίσαμε πάνω από 1.400 περιπτώσεις και ήδη έχουμε ξεπεράσει τις 700 και είμαι βέβαιος ότι και φέτος θα ξεπεράσουμε ε, τις 1500 περιπτώσεις. Ε, στη συνέχεια εδώ σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε την κατανομή κατά εγκλήματα προτεραιότητας. Το βασικό ε, για το Λουξεμβούργο, όχι για τη Eurojust διορθώνει ο μιλητής είναι το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ένα μέρος του συνδυάζεται, τουλάχιστον τα δύο τρίτα συνδέονται και με το οργανωμένο έγκλημα. Το ίδιο ισχύει και ε, με το δουλεμπόριο, το τράφικινγκ, ε, το ξέπλυμα χρήματος και επίσης κοιτάξτε και την τελευταία στήλη παρακαλώ που είναι άλλες περιπτώσεις, ε, υποθέσεις που συνδέονται όμως πάντα με το οργανωμένο έγκλημα. 26 περιπτώσεις ε, μας απασχόλησαν πέρσι σε σχέση με τη διαφθορά. 19 ήταν οι συναντήσεις συντονισμού και δημιουργήθηκε και μια μεικτή ομάδα ε, τότε σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα χρήματος είναι θέμα που σας ενδιαφέρει και εσάς 122 ήταν οι περιπτώσεις πέρυσι για μας είναι ε, το τέταρτο σε σειρά έγκλημα από πλευράς συχνότητας, 27 συνεδριάσεις συντονισμού, δύο μικτές ομάδες έρευνας δημιουργήσαμε και άλλες δύο ε, που συνδέονται με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Και γενικά ε, για το οργανωμένο έγκλημα το 11 είχαμε 197 περιπτώσεις καταγράψει, μόνο για το 11, ε, Ακολούθησαν 56 συνεδριάσεις συντονισμού και 6 μικτές ερευνητικές ομάδες συστάθηκαν. Λοιπόν, τώρα, αν μου επιτρέπετε να σας παρουσιάσω μια συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος μου τελειώνει. Για να σας δείξω και τους περιορισμούς που γνωρίζουμε και τα όρια μας προς το παρόν. Ήταν μια επιχείρηση που την ονομάσαμε επιχείρηση Δράκουλα. Τα πραγματικά περιστατικά. Ήταν ρουμανική η εγκληματική οργάνωση, η οποία είχε εξειδικευτεί μεταξύ άλλων σε ληστείες σε τα κτίρια με εταιρείε με τριπλό α ή πολυεθνικές. Και μόλι είχαν εγκαταστήσει του υπολογιστές, γινόταν ληστεια και τους κλέβανε όλο το ηλεκτρονικό υλικό. Και πώς λειτουργούσαν. Διάλεγαν τα κτίρια όπου ήταν κοντά σε αυτοκινητοδρόμους για να μπορούν να διαφεύγουν εύκολα και γρήγορα και να μεταφέρουν και τα κλοπημαία. Στη Γαλλία, στο Λουξεμβούργο και στο Βέλγιο δραστηριοποιούνταν, αλλά υπήρχαν και διακλαδώσεις στη Δανία, στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα κλοπημαία ε, τα μετέφεραν και τα αποθήκευαν στη Γερμανία, στη συνέχεια τα έστελαν στη Ρουμανία, όπου τα πουλούσαν και ξέπλαιναν και το χρήμα. Συνελήφθησαν οι ύποπτοι και κρατήθηκαν στη Γαλλία, στη Γερμανία και στο Βέλγιο και στις κατοχώρες. Ο Νακριτής στο Λουξεμβούργο ζήτησε ε, να γίνει μια συνεδρίαση συντονισμού σε επίπεδο Eurojust όπου ανέκυψαν τα εξή ζητήματα. Βάσει δεδομένων για τα κλοπημαία και τα ε, επιστραφέντα, ή ε, τα ανακτηθέντα καλύτερα, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το υλικό με μια συγκεκριμένη ληστεία και ε, τοποθεσία. Επίσης, βάση δεδομένων για το DNA και τη σήμανση γιατί είχαμε υλικό από το κλοπημέα DNA, γενετικό, αλλά και από ε, αυτό το υλικό ε, θα μπορούσε να συγκριθεί με γενετικό υλικό κρατουμένων. Και επίσης προσωρινές ε, παραδόσεις, κάποιους που είχαν συλληφθεί σε μία από τις χώρες και ζητούσαν ανακριτές να τους ε, ανακρίνουν σε μια άλλη χώρα. Βεβαίως ήταν και το θέμα της σύγκρουση ε, δικαιοδοσιών, ιδιαίτερα ε, σε ό,τι αφορά την αξιόπινη πράξη του οργανωμένου εγκλήματος. Και ένα τελευταίο, χωρίς να είναι αυτό λιγότερο σημαντικό, κατά τη διάρκεια αυτής τη συνεδρία προτάθηκε να συσταθεί το πρώτο ανακριτή, ειδική ομάδα, μεικτή ερευνητική ομάδα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώ δεν, δεν λέω για ποιου λόγους ε, απερίφθη αυτό, αλλά όλα αυτά τα μέτρα απερίφθησαν που ζητούσε ο ανακριτή. Και τώρα ε, έρχομαι στο παρόν νομικό πλαίσιο της Eurojust. Δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα ακόμα και αν εφαρμοζόταν από όλου η νέα απόφαση. Ε, τη Eurojust, γιατί είναι έτσι το νομικό πλαίσιο. Ζητώ συγγνώμη που με ακρηγόρησε, είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε υποδιευθυντά. Ε, και εμείς καθυστερήσαμε, συλλέξαμε καθυστέρηση και ζητώ συγγνώμη για τη βιασύνη μας τώρα. Θέλω να πω ότι μας έδωσαν ένα δεκάλεπτο παραπάνω οι διερμηνείς, όμως θα πρέπει 12 και 40 παρατήτως να σταματήσουμε. Παρακαλώ λοιπόν να τηρήσετε το χρόνο. Η κυρία Ματιό για το ΕΛΚ έχει πρώτη το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Υποδιευθυντή για την παρέμβασή του, την άκουσα ενδιαφέρουσα και μήπως θα ήταν καλό να έχουμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή μαζί σας, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε τις διαφάνειες που μας προσθέσετε το πρωί, να μας στείλετε ηλεκτρονικά στο email, θα ήταν πολύ καλό για μας. Ευχαριστούμε πολύ αναφερθήκατε στις μικτές αυτές ομάδες και την άρνηση που διαπιστώσατε να υπάρχει από κάποιες χώρες που ειρνούντο να σας διαθέσουν τη συνεργασία σε κάποιες περιπτώσεις. Χωρίς να αναφέρετε συγκεκριμένα κάτι μέλη που αρνήθηκαν, θα ήθελα να ξέρω σε ποιες περιπτώσεις αρνούνται τα κράτη να δημιουργήσουν τις μικτές ομάδες. Για ποιους λόγους, για ποια αίτια προβάλλουν, έχουν βάσιμους λόγους. Ε, μήπως θα μπορούσε κάπως να εξελιχθεί η κατάσταση όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ε, ο κ. Κοτσέτα έχει το λόγο για το S&D. Απλή ερώτηση αντιμετωπίζουμε συχνά για το Eurojust είναι το θέμα της πρωτοβουλίας. Η έλλειψη πρωτοβουλίας αυτό περιορίζει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας. Αυτά μπορεί να κάνει το Eurojust. Το Eurojust δραστηριοποιείται μόνο κατόπιν ετήματος των κρατών μελών. Θεωρείτε μήπως θα ήταν αναγκαίο να περάσουμε σε μία ενίσχυση Τη δυνατότητα να κινηθείτε για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή να δώσουμε εξουσίες περισσότερες στο Eurojust, κυρίως να μπορεί να ξεκινά έρευνε στο Eurojust. Να έχει πρωτοβουλία. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, για την Άλτε. Ο κύριος Νιούτον Ντόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Βγάλτε το καπέλο του Eurojust. Μιλήστε σαν Ευρωπαίος πολίτης, ανήσυχος πολίτης Ευρωπαίος. Σήμερα εκπρόσωπος του Όλαφ είπε ότι χρειαζόμαστε ένα Ευρωπαίο εισαγγελέα. Συμφωνείτε? Χωρίς, όχι υπό την ιδιότητά σας εκπροσώπου αντι, ε, υποδιευθυντού του Eurojust, αλλά σαν πολίτης. Ποια είναι η άποψή σας? Ευχαριστώ. Για την ΚΟΕ, ο κ. Σόντεργκάρ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνατε. Θέσατε το θέμα των δια... της διαφοράς μεταξύ Europol που συλλέγει τις πληροφορίες και του Eurojust που έχει περισσότερο επιχειρησιακό χαρακτήρα. Το πρόβλημά μας είναι ότι επανειλημμένα σε ακροάσεις, σε μελέτες, σε συζητήσεις ακούμε να λέγεται ότι υπάρχουν δυσκολίες, προβλήματα όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ Eurojust και Europol. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Ίσως υπάρχει ένα πρόβλημα με την όλη δομή και ίσως γι' αυτό να υπάρχουν τα προβλήματα συνεργασίας. Ίσως υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο με τον οποίο έχουν δομηθεί οι δύο φορείς. Ίσως υπάρχει πρόβλημα στις εντολές που έχουν δοθεί. Ίσως γι' αυτό να υπάρχουν τα και τα προβλήματα. Θα μπορούσατε να το ξεκαθαρίσετε. Δεν ξέρω αν ισχύει, θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε. Στον κύριο Γιακολίνο, δυνατό τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μας περιέγραψε εκπρόσωπος του Eurojust ποια είναι τα όρια, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των δράσεων του Eurojust. Θα μπορούσατε να μιλήσετε και το ρόλο και για των διαφόρων ε, δικαστικών ε, αρμοδίων για τις επαφές αυτών που διαθέτουν τα κράτη-μέλη για το συντονισμό των ερευνών. Πώς μπορεί να ενισχυθεί αυτός ο συντονισμός, αυτή η συνεργασία μέσω του πιο ενδεδειγμένου της πιο ενδεδειγμένης χρήσης αυτών των σημαντικών ειδικών, αυτών των ανθρωπίνων πόρων, σε ένα πλαίσιο που απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση, κυρίως μεγάλες ικανότητες, μεγάλες επιδεξιότητες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τελευταία παρέμβαση. Ο κύριος Μπορσελίνο, η κυρία Μπορσελίνο έχει το λόγο, συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκπρόσωπος του Τζοστ μας εξήγησε πολύ καλά τι κάνει το Eurojust και τι έκανε. Μας έδωσε και παραδείγματα εξαντλητικά. Εγώ θα σας ρωτούσα τι λείπει από το Eurojust. Ποια είναι τα μέσα που θα θέλατε να διαθέτετε και μέχρι τώρα δεν είχα διαθεσή σας πέρα από αυτά όπω είναι οι μικτές ερευνητικές ομάδες. Το ίδιο θέμα, το ίδιο ερώτησα και τον εκπρόσωπο της Europol και δεν απάντησε. Ε, δεν λειτουργεί λειτουργούν και λόγω, υπάρχουν προβλήματα λόγω ελλείψης χρημάτων, όχι μόνο λόγω ελλείψης εργασίας κάποιων κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά, τα τεράστια που αφαιρούνται από τις χώρες λόγω της παρουσίας του οργανωμένου εγκλήματος, νομίζω ότι δεν κάνουμε σωστά τους υπολογισμούς μας όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι τα μέσα που θα θέλατε να διαθέτετε για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, που όμως μέχρι τώρα δεν είχατε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Δίνω εκ νέου το λόγο στον κύριο Αντιπρόεδρο για ένα πεντάλεπτο για να μπορέσει να μας απαντήσει. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω να αναγνωρίζετε ότι πέντε λεπτά για έξι ερωτήσεις δεν είναι πολύ χρόνο. Το πρώτο ερώτημα ήταν για ποιους λόγους αρνούνται κάποια κράτη-μέλη να ανταποκριθούν στο αίτημα που βάλετε στη συνεδρία συντονισμού για τη δημιουργία μικτής ομάδας. Διάφοροι λόγοι υπήρξαν. Καμιά φορά ήταν βάσιμοι λόγοι. Αυτό που συναντήσαμε χωρίς κατονομάσουμε κάποια χώρα είναι και το εξής. Φόβος. Όσον αφορά τη διεθνή διάσταση ε, είναι κάτι που εμποδίζει μια χώρα να συμμετάσχει στη συνεργασία αυτή και να διαμορφώσει μια μεικτή ομάδα και οικονομικοί λόγοι βέβαια έχουν επιπλέον ε, προβληθεί. Τι εννοώ με τον φόβο της διεθνούς διαστάσεως. Για έναν υπεύθυνο του χώρου είναι σαφές ότι θα πρέπει να κινηθούν δικαστές από την αριστερά πλευρά να βάλουν την υπόθεση δικαστές στη δεξιά μεριά του γραφείου τους. Όταν υπάρχουν υποκράτηση κάποιοι Κρατούμενη προφυλάκηση. Υπάρχει ο κίνδυνος της μακράς προφυλάκησης και πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Και συχνά περιπλέκεται μια υπόθεση με την διαμόρφωση μιας μεικτής ομάδας και φοβούνται ότι λόγω της επιπλοκής αυτής δεν θα μπορέσει να εγκαίρως να ολοκληρωθεί η δίωξη, η υπόθεση. Θεμητός αυτός ο λόγος, κατά την άποψή μου, αλλά θα μπορούσε να προσθέσει ο δικαστης δυο δύο-τρία χρόνια ε, στην ποινή, λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι διεθνής εγκληματική οργάνωση που κινείται διεθνώς. Παρόλο αυτό που δεν έχει διερευνηθεί. Πλήρως. Δεύτερη ερώτηση ήταν η έλλειψη δυνατότητας αναλήψεως πρωτοβουλίας για έρευνες και για διώξεις. Η απάντηση είναι στο άρθρο 85 της ε, συνθήκης της Λισαβόνας που προβλέπει ότι το Eurojust θα εδύνατο να αποφασίσει την εκκίνηση ερευνών και να προτείνει την έναρξη δίω, άσκησης δίωξης. Ετέθη ένα ερώτημα όσον αφορά τη σχέση Eurojust με Europol. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θεμελιώδες πρόβλημα μεταξύ των δύο οργανισμών. Κινούμεθα προς σωστή κατεύθυνση. Δημιουργήθηκαν και μέσα επικοινωνίας. Έπρεπε να επιληθούν διάφορα ζητήματα. Πότε δίνει το Europol πληροφορίες στην Eurojust και τι μπορεί να κάνει το Eurojust. Δίνεται σε εθνικό μέλος, δίνεται στο σώμα, στον οργανισμό, σε άλλο φορέα. Οι πληροφορίες μπορούν να προωθηθούν στις εθνικές αρχές. Όλα αυτά τα ζητήματα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Δεν βλέπω να υπάρχει θεμελιώδες πρόβλημα όσον αφορά την δομή ή τις διαφορετικές δομές που υπάρχουν στο νέο οργανισμό. Η τελευταία ερώτηση ποια ήτανε, τι μπορεί να βελτιωθεί. Συνοψίζοντας, η νέα απόφαση για το Eurojust θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη και βέβαια πιστεύω ότι επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα υπάρξει σχέδιο κανονισμού του χρόνου που θα προταθεί. Κάτι στα πλαίσια του άρθρου 85 ελπίζω. Δεν μιλώ εκ μέρους του Eurojust εδώ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ελπίζω όσον αφορά τι εξουσίε του Eurojust να ισχύει και αυτό. Και η τελευταία απάντηση ζητήθηκε να απαντήσω υπό την ιδιότητά μου ως Ευρωπαίος πολίτης και όχι εν ονόματι του Eurojust. Μπορώ να απαντήσω ότι αυτή η περιπτώση ότι χρειαζόμαστε τον Ευρωπαίο εισαγγελέα διότι τα κράτη-μέλη διαφέρουν πολύ στην άποψή τους για το θέμα αυτό. Αν ρωτήσετε τον Ευρωπαίο πολίτη αυτό είναι πεπισμένο ότι χρειάζεται ένας Ευρωπαίος εισαγγελέα. Ίσως όχι μόνο περιορίζοντα τα συμφέροντά του στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωση σε πρώτη φάση, αλλά ίσως μετά να περάσει και σε άλλη φάση και να επιληφθεί και τη καταπολεμήσεω του οργανωμένου εγκλημάτου. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε Τζέλε, ευχαριστώ κυρίω διότι περιοριστήκατε χρονικά όσον αφορά τι απαντήσει σας. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες δυνατότητες για να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ τους διερμηνείς για την καλοσύνη τους που εργάστηκαν παραπάνω. Διακόπτουμε και συνεχίσουμε τις ακροάσεις αργότερα στις 3 με τον Ιταλό ε, εισαγγελέα τον κύριο Γκράσο θα συνεχίσουμε. Λοιπόν διακόπτουμε εδώ, στις 3 θα ξαναλέμε. Καλή όρεξη.